Καλημέρα σας. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στην ε, συνάντηση της Επιτροπής μας Διεθνούς Εμπορίου. Ο πρώτος Μορέιρα δεν θα προεδρεύσει σήμερα, τουλάχιστον σήμερα το πρωί όχι. Εγώ θα προεδρεύσω, ε, σε πολλά συναδέλφου Στάρντι θα αντικαταθώ σήμερα το απόγευμα. Στα πλαίσια των στόχων ακριβώς να δείξουμε ότι η Ευρώπη είναι η δημοκρατία και ότι μας χαρακτηρίζει η διαφάνεια, η συνάντηση αυτή μεταδίδεται μέσω webstream και να είσαστε και σοβαροί και υπεύθυνοι και χαμογελαστοί. Είναι κατοθετικό η δημοκρατία να δείχνετε ενθουσιασμό όταν λαμβάνετε το λόγο. Πάμε τώρα στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Η κυρία Μουσκαρντίνη σήμερα είναι πουσα. Θα έπρεπε να εξετάσουμε το σημείο για την αξής ε, βάμβακος, την αλυσίδα αυτή και θα το κάνουμε στην επόμενη συνεδρίασή μας και παρακαλώ σημειώστε κάτι ότι θα συζητήσουμε με την ε, αντιπροσωπεία της Επιτροπής ε, της Νέας Ζηλανδίας, ε, εμπόριο, άμυνα κλπ. Και στις τρεις λοιπόν, ε, αλλαγή στην ημερησιά διάταξη, θα συζητήσουμε με την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου της Νέας Ζηλανδίας στις 3 το απόγευμα και έτσι θα είμαστε και σίγουροι ότι στις 4 θα διεξαχθεί η ψηφοφορία μας. Το σημείο 2, αφού πρώτα μου πείτε ότι συμφωνείτε με την αλλαγή της ημερήσιας διάταξης. Εντάξει, εντάξει. Δεύτερο, έγκριση των πρακτικών της συνεδρίας της 17ης και 18ης Σεπτεμβρίου 2012. Εγκρίνονται. Κανένα σχόλιο, καμία αντίρρηση τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σημερινής πρωινής μας συνάντησης. Ε, το σημείο 3 τώρα τους φακέλους σας ε, έχετε όπως συνήθως τα σημεία που έχουν να κάνουν με τις ανακοινώσεις του Προέδρου και αν θέλετε να δείτε, κοιτάξτε το φάκελό σας. Διαφορετικά, αν έχετε κάτι να ρωτήσετε ειδικό, θα το συζητήσετε με τον Πρόεδρο. Το σημείο 4 τώρα. Εδώ στο σημείο 4 Έχουμε τις συμφωνίες ε, για τις επενδυτικές μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών και τις μεταβατικές ρυθμίσεις. Ο προς Μορέιρα ασχολείται με το θέμα αυτό. Και σε ποια φάση βρισκόμαστε σε αρκετά ενδιαφέρουσα της όλης διαδικασίας ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Προχωράμε στη μελέτη των θέσεων του Συμβουλίου μετά από την πρώτη ανάγνωση, το Συμβούλιο θέτησε τις 4 Οκτωβρίου την θέση του και ο κ. Μορέιρα ε, δεν μπορεί να έρθει εδώ σήμερα, αλλά σίγουρα θα συνεχίσει την εργασία του πάνω σε αυτό το θέμα. Και δεν ξέρω μήπως υπάρχει κάποια αντίρρηση ανάμεσά σας. Ε, κανονικά ο κύριος Μορέιρα θα πρέπει να συνεχίσει αυτό το θέμα στα πλαίσια και της προοπτικής της δεύτερης ανάγνωσης. Το Μπέτλονγκερ θα ακούθησετε σήμερα γιατί αντικαθιστά επίλεκτο μέλος, ε, ακριβώς ε, αντικαθιστά τον πρόεδρο Μορέιρα που θα μας πει ένα πράγματα εκ μέρους του πρόεδρου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Φυσικά δεν μπορώ να τον αντικαταστήσω, αλλά μπορώ να μοιραστώ κάποιες ιδέες που μου κοινοποίησα σχετικά με την έκθεση αυτή. Είχαμε λοιπόν τον τριμερή διάλογο με συμφωνία στην οποία καταλήξαμε το Μάιο φέτος από την οποία Στη συνέχεια έστειλε στο κορεπέρο ο κύριος Μωρήρα ένα κείμενο, μια επιστολή, για να ρωτήσει αν μπορεί το κείμενο αυτό να γίνει δεκτό και από το Συμβούλιο. ώστε να προχωρήσει χωρίς δεύτερη ανάγνωση από το Κοινοβούλιο. Κάποια θέματα νομικού, νομοτεχνικού χαρακτήρα χρειάστηκε να κρυθούν. μέχρι να υιοθετήσει το Κοινοβούλιο το έγγραφο αυτό. Ο κύριος Μωρέιρα τα δέχτηκε ως νομοτεχνικά ζητήματα και όχι ουσιαστικής ε, σημασίας. Και έτσι προτείνει να επικυρώσουμε χωρίς τροπολογίες την απόφαση του Μαΐου. Αυτή είναι η σύσταση, την έχετε στην αεροφάση σας και ως εκ τούτου στο πλαίσιο της δεύτερης ανάγνωσης έχουμε τρεις μήνες στη θέση μας, μέχρι τον Ιανουάριο πρέπει να εγκριθεί, αλλά για να είμαστε και σίγουροι ας τη φέρουμε καλύτερα στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. Για να δω τους κοιόδης εισηγητές. Δεν είναι ο συνάδελφος. Α, την ε, σφιλελεύθερος δεν είναι. Φρανσίσκα Κέλλερ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λάγκε. Νομίζω ότι ήταν ε, δύσκολη ε, εμπειρία αυτή για μας, ε, αυτό το έγγραφο. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Μορέρα και τους υπόλοιπους και ισχυτές και τον κύριο Ζαλεύσκη όλος ιδιαίτερος για την αποφασιστικότητά τους ε, καθ' όλη τη διαδικασία. Θα θυμάστε ότι οι πράσινοι ε, συμμετείχαν πολύ ενεργά σε αυτό το θέμα. Οι βάσεις ε, προήλθαν από το εισηγητή μας, τον Κάρος Λούτε που ήταν ο πρώτος εισηγητής για το θέμα αυτό και στη συνέχεια χρειάστηκε να υπαναχωρήσουμε, να παρετηθούμε, επειδή πρότεινε μία ρήτρα εκπνοής. νομίζω ότι οι περισσότεροι πιστεύουν ότι θα έπρεπε η θέση του Συμβουλίου να ε, ενταχθεί ε, να εγκριθεί ε, και να την ενσωματώσουμε και εμείς μάλιστα στη δική μας θέση. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό. Νομίζω ότι έχει παρέλθει λόγω των εξελίξεων. Επειδή έχουμε κάποια θεσμικά προνόμια και λόγω των νέων αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου στην επενδυτική πολιτική, Αυτό είναι κάτι το οποίο βέβαια έθεσαν αμφιβόλο κάποιες ε, δυνάμεις του ε, Συμβουλίου. Πρέπει να δούμε το γεγονός ότι είναι πολύ, ε, δεν είναι καθόλου ικανοποιητική η κατάσταση της νομοθεσίας που αφορά συγκεκριμένα αυτό το θέμα γιατί βρισκόμαστε σε μια μεταβατική διαδικασία. Είμαστε στην διάρκεια της ολοκλήρωσης μεταβατικής διαδικασίας για την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην επενδυτική πολιτική. Δεν υπάρχει καμία όμως ε, βεβαιότητα ότι όντως θα γίνει αυτό στο μέλλον και ότι η ε, αποκλειστική δυνατότητα των κρατών μελών να αποφασίζουν γι' αυτό θα είναι πλέον ε, στο παρελθόν. Εμείς έχουμε σκοπό λοιπόν να καταψηφίσουμε τη συγκεκριμένη νομοθεσία ως πράσινη και ελπίζω να το αποδεχθείτε αυτό μετά από όλη τη δουλειά που κάναμε για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Χέλμουτ, λέει ο ε, Κύριο Σόλτς, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ σε κάποιε ιδέε και προτάσει τη ομάδα μα σε σχέση με τη συμφωνία αυτή, χωρί να επισέλθω στο ιστορικό τη εξέλιξη όλη αυτή τη υπόθεση. Γιατί έχει γίνει μακρά ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή μα. Έχουν ακουστεί διαφορετικέ προσεγγίσεις και θα ήθελα και εγώ να υπογραμμίσω ότι δεν είναι ικανοποιημένη με τα αποτελέσματα η ομάδα μας. Πάντως σεβόμαστε τη σκληρή δουλειά, δουλειά που έκανε η ομάδα των αντιπραγματεύσεων για τον τριμερή διάλογο. Αναγνωρίσουμε ότι επιτάπητος αυτή τη στιγμή βρίσκεται ότι περισσότερο θα μπορούσε να εξασφαλίσει από τις θέσεις του το Κοινοβούλιο σε σχέση με την αρχική θέση με την αρχική πρόταση, όπως υπεγράμμισε και η κυρία Κέλλερ τώρα. Ίσως είδαμε πολύ πρόωρα το πού θα μπορούσε να εστιαστεί ο συμβασμό. Γι' αυτό λοιπόν θα περιμένουμε και το τελευταίο γύρο των διαπραγματεύσεων για να τοποθετηθεί η ομάδα μας, όσο όχι τόσο ριζοσπαστικό, τόσο ριζικά όσο αυτό που είπε η Σκακέλλερ. Αλλά πάντως περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει στις τελικές διαπραγματεύσεις και πρέπει να ομολογήσω ότι διστάζουμε ως προς το ναι για το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να πείσει το συνάδελφο πάνω στο θέμα αυτό, τον κύριο Σόλτ. Όχι. Από την Κυπριακή Προεδρία κάποιος θα επιθυμούσε το λόγο παρακαλώ για την ε, θέση του Συμβουλίου. Όχι. Δεν βλέπω κανένα. Εκπρόσωπος της Επιτροπής τότε. Ο κ. Ρουμπινάτσι. Παλασίε Σουρέιντα. Βεσγκρινς κάπως έτσι. Ε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Η Μάρτα Μπούς από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η Επιτροπή ενέκρινε τη θέση της ε, σε σχέση με την θέση του Συμβουλίου κατόπιν πρώτης ανάγνωσης και στην ανακοίνωσή της, της 16 Οκτωβρίου του 2012, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωση αυτή επιβεβαιώνει σαφώς ε, την θέση ε, του Συμβουλίου στην πρώτη ανάγνωση, επιβεβαιώνοντας ότι η θέση αυτή αντικατοπτρίζει πλήρως την συμφωνία ε, που συνήφθη στις τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Συνεπώς, το, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται τη θέση ε, του Συμβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για όσα μας ενημερώσετε. Αλλά ε, άλλαξε η γαλλική διερμηνία αντί για το 3 είναι στο 2 κανάλι. Μπέρντ Λάγκε. Μπέρντ. Ευχαριστώ πολύ. Αντιλαμβάνομαι ότι οι συνάδελφοι παραμένουν επιφυλακτικοί και φαίνεται ότι εντωμεταξύ αρκετά κράτη-μέλη έχουν αναγνωρίσει ότι και η εμπορική πολιτική και η προστασία των επενδύσεων, σχετική συμφωνία δηλαδή, έχουν ε, σημαντικό ρόλο ανοίξει για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν, εάν κανείς ε, κοιτάξει με μια στάση αφιψηλού την ε, κατάσταση ε, μπορεί να, μπορεί να θεωρήσει ότι θα μπορούσαμε να είχαμε επιτύχει πολύ περισσότερα πράγματα. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι είναι πολύ καλή η συμφωνία. Έχουν γίνει... Ε, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα και νομίζω ότι η συμφωνία μπορεί να περάσει έτσι. Σας ευχαριστώ. 9 Νοεμβρίου μεσημέρι για τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Σημείο 5 τώρα. Πώς έχουν, ε, σε ποιο στάδιο είναι οι διαπραγματεύσεις για τον τριμερή διάλογο, τις διαπραγματεύσεις στη δεύτερη ανάγνωση για τη μακροοικονομική βοήθεια στη γεωργία. Δυστυχώ είναι απόν όπω είπαμε ο πρόεδρο Μορέιρα. Άρα λοιπόν ο Μπέρτ Λάγκε έχει το λόγο που τον αντικαθιστά υποχρεωτικά. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ συνάδελφοι. Ο Βιτάλ Μορέιρα είναι εισηγητή για την έκθεση. Και μου είπε ότι πρέπει να σας ενημερώσω πως στις 16 Οκτωβρίου έλαβε χώρα ένας πρώτος τριμερής διάλογος όπου ιδιαίτερως συστήθηκαν οι δυνατότητες για μια μεσοπρόθεσμη λύση, ενδιάμεση λύση. προκειμένου να απεμπλακεί η κατάσταση, χωρίς όμως αποτέλεσμα δεν εξασφαλίστηκε συμφωνία με το Συμβούλιο και ειδικότερα και εδώ πάλι τα κρατη δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν μια, ε, με ενιαίο τρόπο το, τη θέση του Κοινοβουλίου. Έτσι λοιπόν. Τα κράτη-μέλη στο εσωτερικό τους, στην ομάδα τους προσπαθούν να αναζητήσουν λύσεις και δυνατότητες απεμπλοκής της κατάστασης και μάλλον θα, μας, θα είναι έτοιμα την επόμενη εβδομάδα. Φαντάζομαι ότι θα γίνει νέος τριμερής διάλογος στη συνέχεια. Ωστόσο δεν έχει οριστεί ακόμη η ημερομηνία του προσεχούς, της προσεχούς συναντήσεως. Και έτσι συνεχίζουμε με την τυπική διαδικασία και πάμε στη δεύτερη ανάγνωση. Αναλόγως δεν ψηφίζουμε. Ο πρόεδρος κάποιο σχόλιο από άλλα μέλη. Γκάρντα από το ΕΛΚ. Κανείς. Τίποτα. Μήπως θα ήθελα να λάβει το λόγο η Επιτροπή. Αρούνας Ριμπόκας. Oui. Thank you, Chairman. Ε, Ευχαριστώ. Είμαι εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου και δεν είναι δική μας αρμοδιότητα αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Για να δούμε. Τη σύσταση του εισηγητού να την υιοθετήσουμε, να πάμε στη δεύτερη ανάγνωση. Το Δεκέμβριο λύνει η προθεσμία οπωσδήποτε για μια συμφωνία. Διαφορετικά χρειάζεται να πάμε στην επόμενη φάση. Χωρίς μικρόφωνο, πρόεδρος, δεν ακούμε. Χωρίς μικρόφωνο. Το σημείο 6. Δραστηριότητες εποπτικής ομάδας. Κύριος Καμάλ απόλ. Είτε θα το δούμε σε λίγο, είτε μήπω κάποιο άλλος θα ήθελε να πει μερικά πράγματα για τη Σιγκαπούρη και για τη συνάντηση με τον πρέσβη της Σιγκαπούρης. Όχι, κανείς. Να πάμε στην Κίνα τότε. Ο Γκώδης, φάκελος, ε, σοβαρό θέμα για την Ευρώπη. 17 Οκτωβρίου συνάντηση πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στη Γενική Διευθυνσία του Εμπορίου και του Ανταγωνισμού της Επιτροπής τον Χέλμουντ Σόλτς να ακούσουμε για την επικαιρότητα για την Κίνα και έλεγα ο Γκόδη Φάκελος ε, γιατί διεξάγει έρευνα τη Γενική Διεύθυνση για τα φωτοβολταϊκά και για το ντάμπινγκ και τα όσα έχει αναγγείλει η Κίνα μόλις χθες και για αντίπεινα. Γιατί ξεκινάει η έρευνα για ντάμπιν, για από τα υλικά που κατασκευάζονται τα φωτοβολταϊκά. Ο Χέλμουντ Σόλτς. Ευχαριστώ πολύ. Και οι, και οι πράσινοι έχουν ε, συμβάλλει στη διατύπωση αυτής της ε, πρότασης για τα φωτοβολταϊκά. Θα ήθελα πάντως να αναφερθώ στην τελευταία συνεδρίαση για, την, ε, για τη σχέση με την Κίνα, όπου συζητήσαμε θέματα της ε, τελευταίας συνόδου κορυφής του Σεπτεμβρίου. Θέματα ενδιαφέροντα και ευαίσθητου χαρακτήρα στη σχέση μας με την Κίνα. Και κοιτάμε και τα θέματα της ε, τελευταίας, ε, του τελευταίου μνημονίου συνεννόησης με την Κίνα για τα θέματα του αγωνισμού. Ενημερώνω λοιπόν τους συναδέλφους ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 20 Σεπτεμβρίου υπέγραψε μνημόνιο συνεννόησης με την Κίνα, το οποίο περιλαμβάνει, ορίζει ένα πλαίσιο για τη συνεργασία και πάνω απ' όλο το συντονισμό μεταξύ αφενός Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφετέρου της αρχής μονοπωλίων της, της Κίνας και της ε, Επιτροπής για τις, ε, πολιτικές, ε, για τις μεταρρυθμίσεις στο εμπόριο, στο διεθνές εμπόριο της κινέζικης κυβέρνησης και αντίστοιχα της ομάδας για το εμπόριο και τη βιομηχανία της Κίνας. Άρα λοιπόν εξετάστηκε εκεί καλύπτεται μάλλον η νομοθεσία, η υλοποίηση της εφαρμογή της και η τεχνική συνεργασία γύρω από τα θέματα της, των καρτέλ καθώς και μηχανισμοί άμυνας για την αντιμετώπιση προβλημάτων ε, δεσπόζουσας θέσης. Στη δε συνεδρίαση αυτή της ομάδας αποπτίας, στη συζήτηση, και θα ήθελα και επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω, έστω και αν ε, δεν ε, είναι όλοι οι συνάδελφοι μέλη της εποπτικής ομάδας, συμμετέχουν όλες οι ομάδες και η γραμματεία πάνω απ' όλα. Θέλω λοιπόν να ευχαριστώ για την ε, συμμετοχή και τη συνδρομή. Το θέμα της μετάβασης συζητήθηκε πώς μπορούμε να το επιλύσουμε. Ειδικότερα το ζήτημα των διμερών σχέσεων σε επίπεδο εμπορικό ανταγωνισμού, βιομηχανικής συνεργασίας. Πώς μπορεί να ενισχυθεί αυτή η σχέση και τι είδους εξελίξεις μπορούμε να περιμένουμε από το ε, συνέδριο του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος που θα γίνει σύντομα ως προς την νομοθεσία αυτή, όπως επίσης και τι είδους επιρροή μπορεί να έχουν αυτές οι αποφάσεις του συνεδρίου του Κινέζικου Κομμουνιστικού κόμματο, προς την πολιτική της χώρας. Ήταν μια ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων με τον ε, Πρωθυπουργό Βεντζαμπάου ως προς τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη μετάβαση της Κίνας σε μια οικονομία αγορά. καθώς και το ζήτημα των ε, διμερών σχέσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δε εκπροσωπείται με ύψη, σε στο επίπεδο από τον Επίτροπο Ντεγκούχτ σηματοδοτώντας τη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οικονομική συνεργασία με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Επίσης, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημειώνουμε ότι έκανε κάποιες διαπιστώσεις σχετικές με την ε, ε, λειτουργία και την παρουσία του γραφείου για τις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα που βρίσκεται στο Πεκίνο, ότι ε, σημειώνεται από εκεί πολύ θετική εξέλιξη στο κλίμα. Παραμένουν βέβαια προβλήματα προς την πρόσβαση στην αγορά. Και εδώ, μου επιτρέπετε, θα ήθελα να κάνω μια προσωπική παρατήρηση ότι ίσως θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξανασυζητήσει ακριβώ τι σημαίνει πρόσβαση στην αγορά. Τι σημαίνει για μα πρόσβαση στην αγορά επ' τι οικονομικέ συνθήκε όταν έχουμε να κάνουμε τόσο ισχυρέ οικονομικά χώρε και αγορέ, όπω η Κίνα. Αλλά δεν αφορά μόνο την Κίνα, αφορά γενικότερα και άλλα κράτη Αυτό αυτός ο προβληματισμό Ινδία, Βραζιλία ή και Μερκοσούρ εν γέννη. Φερρυπίν, πρέπει εμεί για μα να ορίσουμε τι εννοούμε όταν λέμε πρόσβαση στην αγορά. Ίσως χρειαστούν νέοι ορισμοί. Η νέα αντίληψη και συναντήληψη αυτών των ενιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. έτσι ώστε να ε, μπορούμε να συζητήσουμε συνθήκες ε, εμπορικών σχέσεων, συναλλαγών, πόρους, ισότιμους, δίκαιους, θεμητούς με τους εταίρους μας. Ξέρουμε επίσης ότι οι Κινέζοι ενδιαφέρονται για περισσότερα βήματα και διμερείς συμφωνίες εμπορικών συναλλαγών που να καλύπτουν περισσότερους τομείς. Και πρέπει ίσως να το σκεφτούμε αυτό πιο σοβαρά. Ίσως είναι νωρίς ακόμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά εάν έχουμε με άλλους εταίρους της, διεθνούς, ε, της παγκόσμιας κοινής ε, ήδη τέτοιου είδους ε, επαφές, θα έπρεπε ίσω και ο Γιάννη το επισήμανε νωρίτερα να εξετάσουμε πιο προσεκτικά τι είδου σχέσει μπορούν να έχουν επιχειρήσει μεταξύ του σε συγκεκριμένου τομεί, όπω για παράδειγμα τη ηλιακή ενέργεια ή η αιωλική που θα είναι το επόμενο θέμα. Ε, Πώ δηλαδή μπορεί το θέμα, το ζήτημα των ε, πλεονεκτημάτων που μπορεί να προσφέρει μια ευρωπαϊκή επιχείρηση ως προς την ε, εφαρμοσμένη έρευνα, την τεχνολογική εφαρμογή, τη βιομηχανική παραγωγή να προσφέρουν και ταυτόχρονα πώς μπορεί να υλοποιηθεί μια μαζική παραγωγή σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις ε, στην Κίνα ή όπως είπα και σε, άλλα τρίτα κράτη. Τόσο προς όφελος των πολιτών, όσο και γιατί δεν πρέπει να το λησμονούμε, έχει πολύ σημαντικό ρόλο όσο και αν παραγνωρίζεται μερικές φορές ε, για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Και θα πρέπει να κάνουμε προσπάθεια στην κατεύθυνση αυτή. Και έτσι λοιπόν αυτή η διμερή σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας μπορεί να έχει μεγάλη σημασία. Δεν πρέπει να χάσουμε την προοπτική αυτών των σχέσεων και βέβαια των μεγάλων προκλήσεων στις ε, σχέσεις μας ε, με τους μεγάλους εταίρους. Επίσης κάτι άλλο που δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε είναι το θέμα της ε, συμμετοχής της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Τα τελευταία 15 χρόνια τι έχει γίνει με την παρουσία της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, τι δεν έχει γίνει. Είναι όλα θέματα τα οποία πιστεύω χρειάζεται να συζητήσουμε και υπό το φως των αποτελεσμάτων ε, της ε, κοινοβουλευτικής συνέλευσης ε, της, του ΠΟΕ που θα λάβει χώρα την προσεχή εβδομάδα. Και άρα καλό θα είναι να τα δούμε όλα αυτά μαζί, να δούμε πώς και άλλα όργανα και μάλιστα πολυμερούς συνεργασίες επίσης ή από την άλλη συζητούν και διαπραγματεύονται τα θέματα αυτά και πώς ενσωματώνουν τις εμπορικές πτυχές μιας συνεργασίας στα ε, στι συζητήσει του, έτσι να δούμε και εμεί πώ μπορούμε να συμβάλλουμε και να ενισχύσουμε ή να, να υπογραμμίσουμε τι θέσει Ευρωπαϊκή Ένωση αυτέ τι πολυμερεί διαπραγματεύσει. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Κάποιο σχόλιο, μήπω ε, κάτι θα θέλατε να προσθέσετε, Όχι. Εγώ όμω κάτι θα ήθελα να προσθέσω. Ο Ρίγμουντ Σόλτ ε, μίλησε για τα φωτοβολταϊκά είναι κάτι το εμβληματικό της όλης καταστάσεως για τις εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα. Γιατί εμβληματικό. Βλέπουμε μια τεράστια χώρα, την Κίνα, με βιομηχανική τεράστια δυνατότητα που πιστεύει ότι οι ανανόσιμες ενέργειες στρατηγικά είναι ουσιαστικό σημείο του 21ου αιώνα. Και αφετέρου εγώ δεν είμαι υπέρ ενός σχεδιασμού με το στυλ Κίνας, αλλά αν συγκρίνουμε το πενταετές κινέζικο πρόγραμμα και τα όσα λέμε για τη βιομηχανική πολιτική του αρμόδιου επιτρόπου δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εντάξει, δεν θα ήθελα να έχουμε πενταετές πρόγραμμα στην Ευρώπη. Αλλά αν δεν υπάρχει κάποια σοβαρή φιλοδοξία είτε στη βιομηχανική επιλογή εργαλεία ευρωπαϊκά για να ξέρουμε προς τα πού πηγαίνει η ευρωπαϊκή οικονομία και πώς θα υπερασπίσουμε τα συμφέροντα τα ευρωπαϊκά και τη βιομηχανική μας δυνατότητα και τα συμφέροντα το με αυτό. Σήμερα δεν είμαστε κατάλληλα εξοπλισμένοι σε χώρες απέναντι όπως την Κίνα και πώς θα συνδυαστεί η βιομηχανική μας πολιτική με την υπόλοιπη δεν έχουμε τα καταλόπλα. Βλέπουμε ότι η Κίνα οικοδόμησε τις σχέσεις ε, σε πολλαπλό επίπεδο, περισσότερο με κάθε κράτος ε, ξεχωριστά από την Ευρώπη παρά μόνο όλη την Ευρώπη για να μην υπάρχει μια ισχυρή θέση της Ευρώπης στην εμπορική πτυχή κυρίως. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που σήμερα δεν έχει τα κατάλληλα βαριά όπλα, έτσι βλέπουμε τα πράγματα στα φωτοβολταϊκά, θα απαιτηθούν μήνες, ενώ υπάρχουν επιχειρήσεις που κλείνουν σήμερα στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν δεν επωφεληθεί από την ευκαιρία αυτή για να δει τις σχέσεις εμπορικές με την Κίνα, ότι είναι της Ευρώπης ολόκληρης και των θεσμικών οργάνων της Ευρώπης, την Επιτροπή, αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, τότε θα επικρατήσει η Κίνα επειδή εμείς δεν θα έχουμε μια συμπληρωματική σχέση με συνοχή επικοδομητική στη σχέση μας με την Κίνα. Άρα λοιπόν είναι σημαντική αυτή η περίοδος και η Ευρώπη δεν θα πρέπει να χάνει το στόχο της. Κυρία Μπρέντερ, Μπέρντερ, Μπέρντερ. Um, Ευχαριστώ πολύ. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι εκτός θέματος αυτό που θα πω, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο πιστεύω ότι θα έπρεπε να θέτουμε κάθε φορά όταν ε, συναντιόμαστε και διαπραγματευόμαστε με τους Κινέζους και αυτό είναι η υποστήριξή τους ε, για το παράνομο εμπόριο ε, στο, σε ελεφαντοστό και κέρα το ρινοκερο. Είναι κάτι το οποίο γίνεται πάρα πολύ καιρό ε, στην Αφρική. Είναι κάτι το οποίο γίνεται με μια σιωπηρή συμφωνία ε, της κυβέρνησης ε, εκεί, γιατί γίνεται παράλληλα με το, ε, με το νόμιμο εμπόριο που γίνεται ε, στα προϊόντα αυτά. Αν καταφέρουμε λοιπόν ε, να σταματήσουμε το dumping στην Ευρώπη για φωτοβολταϊκό εξοπλισμό, το, επόμενο, το επόμενο μέρος στο οποίο θα μετακινηθεί αυτό είναι στην Αφρική. Βλέπουμε ας πούμε τι γίνεται με την Κένια στέλνουν εκεί τον εξοπλισμό, ε, δεν δουλεύει ο εξοπλισμός και τότε ο κόσμος κάνει την όρεξή του να αγοράσει νέο εξοπλισμό. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια ε, ευρύτερη θεώρηση, συνολική θεώρηση όταν μιλάμε με την Κίνα και με άλλες αναδυόμενες μεγάλες αγορές με τις οποίες δεν πραγματευόμαστε γιατί εδώ έχουμε μια αγορά στην οποία θέλουν να έχουν πρόσβαση και αυτό μας δίνει ε, ένα μοχλό πίεσης να ε, ηγηθούμε εμείς και να συζητήσουμε ε, ζητήματα πάρα πολύ σημαντικά και το παράνομο εμπόριο ελεφαντοστού είναι κάτι το οποίο όλο και περισσότερο συμβαίνει στην Αφρική. Πρώτα μα στο χέλμου το λόγο, μήπως κάποιο σχόλιο από πλευράς Επιτροπής. Κανείς η Κίνα, η Επιτροπή σας ενδιαφέρουν ή όχι. Όχι φαίνεται. Ο Χέλμουτ. I guess it is interesting for the Commission, but maybe... Πρέπει να είναι ενδιαφέρον. Πρέπει να είναι ενδιαφέρον για την Επιτροπή, από ό,τι υποψιάζομαι, αλλά μάλλον δεν θέλουν να εκτεθούν εδώ τώρα να κάνουν συζήτηση για το θέμα αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Οι διμερεί εμπορικέ σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Επιτροπή έχουν μεγάλη σημασία. Συμφωνώ στα όσα υπόθηκαν. Απλώ θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιε παρατηρήσει σα. Διότι Από ό,τι βλέπω εγώ την κατάσταση. Αν δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς τι είναι αυτή η αγορά του 1,4 εκατομμυρίων ανθρώπων που είναι οι πολίτες της Κίνας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε και τη σημασία της αγοράς αυτής για τους άλλους εμπορικούς εταίρους της Κίνας, αλλά και τις προκλήσεις που συνεπάγεται αυτή η αγορά για τις πρώτες ύλε, για την παραγωγή, για τα τρόφιμα, για το κλίμα. Άρα λοιπόν, πρέπει και να αναλογιστούμε τι συνέπειε μπορεί να έχει αυτή η μεγάλη αγορά και τι, τι σημαίνει αυτή, αυτό το μέγεθο, αλλά και εμείς τι δικές μας τις ε, σχέσεις και τη συμπεριφορά. Τι κάνουμε. Ίσως λοιπόν δεν έχουμε ακόμη αντιληφθεί τι συνέπειες έχει για μας αυτή η εμπορική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Φέρει στα φωτοβολταϊκά. Για τη Γερμανία τουλάχιστον. Η βιομηχανία των φωτοβολταϊκών στη Γερμανία αποκοιμήθηκε λίγο γιατί δεν επένδυσε σε περαιτέρω επιτάχυνση, σε ανάπτυξη, σε νέες τεχνολογίες. Απλώς εισέπραξε τις επιδοτήσεις, κρατικές επιδοτήσεις και προχώρησε στην παραγωγή. Αυτό δεν μπορεί βέβαια να του δώσει ανταγωνιστική θέση σε σχέση με την αντίστοιχη βιομηχανία φωτοβολταϊκών της Κίνας. Γιατί είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες, οι όροι, οι, οι ιδέες που καθοδηγούν ε, τους χειρισμούς των ανταγωνιστών. Άρα χρειάζεται μια πιο προηγμένη παραγωγή, μια πιο καλά μελετημένη παραγωγή φωτοβολταϊκών. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο αντιμετώπισης. Και, και θα έλεγα επίσης ότι ίσως πρέπει από αυτές τις νέες προκλήσεις να συζητήσουμε και τη στρατηγική 2020 για τις εμπορικές μας σχέσεις, γιατί νομίζω ότι πρέπει να επιταχύνουμε και να δούμε πώς εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με κοινέ προδιαγραφές, με διεθνείς συμφωνίες, με αξιόπιστες συμφωνίες για τις εμπορικές σχέσεις. Και άρα πρέπει νομίζω να ε, καλλιεργήσουμε την ευαισθητοποίηση, να ενισχύσουμε την ευαισθησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις δικές μας ευθύνες, πρώτα στο εσωτερικό της Ένωσης και μετά να ζητούμε από τους εταίρους μας να είναι και αυτοί σωστοί και έντιμοι απέναντί μας. Εντάξει, ευχαριστώ είναι 10% το κόστος μικρότερο. Δεν είναι εκεί η τιμής ε, πάνω στους καθρέφτες των φωτοβολταϊκών 10 ε, δισεκατομμύρια, αλλά δεν υπάρχει και τόση προσπάθεια. Και το απόγευμα το γνωρίζετε ότι θα έχουμε την ακρέαση ένα workshop για τις επενδύσεις στην Κίνα και σίγουρα η Επιτροπή θα έχει κάτι να πει. Μερκοσούρ και Κεντρική Αμερική. Για το Μερκοσούρ έχουμε τον Τζον Λούκας ε, την έκθεση και τον Παύλο Σάλπα οι οποίοι πήγαν μέχρι εκεί και στη Βραζιλία και στην Κοσταρίκα και στον Παναμά. Λοιπόν, ε, να ακούσουμε τα σχόλιά τους ε, για τα ταξίδια τους αυτά, τις εντυπώσεις τους και μετά εάν ο Λάγκε συμφωνεί ίσως να πει μερικά πράγματα για το... Θα έχουμε μια έκθεση για τι ακριβώς ε, σκεφτόμαστε για την Ρωσία, η αντιπροσωπή για τη Ρωσία μετά από τις ε, δύο εισηγήσει που θα ακούσουμε. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι, κύριε Σούστα, σαν εισηγητής ε, συνόδευσα την αντιπροσωπεία στη Βραζιλία και αυτό μετά από ένα γύρο διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ευρώπη και το Μερκοσούρ σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις και την κάπως πιο περίπλοκη συμφωνία σύνδεσης. Έχει προχωρήσει η ώρα και έχουμε πολλή δουλειά σήμερα. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται περισσότερο περιληπτικός. Να σας πω ότι καθαρά φάνηκε ότι είναι το σύστημα σχέσεων ανάμεσα σε εμά και τη Βραζιλία, Βενεζουέλα, Αργεντινή, Ουρουάη και την Παραγουάη παρά το τι ισχύει από εκεί από πολιτικής πλευράς. Είναι λοιπόν μια στρατηγική πολύ σημαντική. Όλα αυτά που θέτουν δυσκολίες σε μια συμφωνία αλλά όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για μας και ισχύει επίσης ότι όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή του κόσμου εκεί και σε σχέση με περισσότερο εμπορικά θέματα και όχι μόνο πολιτικά καθυστερούν σίγουρα την όλη διαδικασία. θα πρέπει να αντιληφθούμε και τι σημαίνει και η είσοδος της Βενεζουέλας στο Μερκοσούρ τώρα πρόσφατα και δόθηκαν και μαθήματα μπορούμε να πούμε με τις εκλογές και θα δούμε τι έγινε με τις εκλογές και όσα συνέβησαν τις προηγούμενες μήνες στην Παραγουάη επιβαρύνει ιδιαίτερα τη σχέση ανάμεσα στις χώρες του Μερκοσούρ και ακόμη κάτι η πολιτική της Αργεντινής για τις εμπορικές σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο χαρακτηρίζονται αυτές οι σχέσεις όλο και περισσότερο από ισχυρό προστατευτισμό και οθεί και απαντήσεις προστατευτισμού από πλευράς και της Βραζιλίας στο όλο παγκόσμιο πλαίσιο. Τα αναφέραμε αυτά και στις αρχές ε, που συναντήσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών της Βραζιλίας και τον Υπουργό Γεωργίας ε, Συναντηθήκαμε επίσης με επιχειρηματικούς κύκλους, με μη κυβερνητικές οργανώσεις και διάφορα σεμινάρια στην, στο Πανεπιστήμιο της, στη Φλωριανόπολη και προσπαθήσαμε να καταλάβουμε την κατάσταση, την πολιτική, με τις εμπορικές σχέσεις και από πλευράς εμπορικών σχέσεων στο σύνολο του κόσμου. Ειδικά αυτό το γύρο διαπραγματεύσεων που μας δείχνει μια κατάσταση. Δεν είναι ότι οπισθοδρομήσαμε, αλλά ταυτόχρονα δεν προχωρήσαμε κιόλας. Ο γύρος των διαπραγματεύσεων μας δίνει να καταλάβουμε το Μερκοσούρ αυτό καθ' αυτό δεν είναι ικανό να παρουσιάσει μια κατάλληλη πλατφόρμα για συζήτηση και για το Σαντιάγκο, για την διάσκεψη κορυφής του Ιανουαρίου θα πρέπει να δούμε τα πράγματα, γι' αυτό από δική μας πλευρά θα πρέπει να συλλογιστούμε καλύτερα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επειδή χρειάζεται εμείς να καταθέσουμε ένα ψήφισμα που να συγκλίνουν οι διάφορες συνιστώσεις, να βλέπουμε τις διάφορες δυσκολίες αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στα πλαίσια του Μερκοσούρ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσεις ε, με διαφορετικές απόψεις, με ένα ψήφισμα που τώρα πια έχει ξεπεραστεί από τα, για τα γεγονότα και ένα ψήφισμα για τα γεωργικά θέματα που ανάγεται στο 2011, είναι παλιό. Είναι δυσκολίες αυτές που δεν τις λάβαμε υπόψη μας ε, Βενεζουέλα, Παραγουάη, προστατευτισμός της Αργεντινής και κάποιο προστατευτισμό από πλευρά Βραζίλια. Γι' αυτό στο Συμβούλιο θα πρέπει να δούμε την εντολή για τι διαπραγματεύσει και επίση από πλευρά Κοινοβουλίου μια κάποια σκέψη για να συνοδεύσει τη συζήτηση στη διάφορα φόρουμ τα ευρωπαϊκά και σε σχέση με τα όσα θα συζητηθούν τον Ιανουάριο στο Σαντιάγκο. Βέβαια δεν είναι ότι έχει κλείσει η πόρτα, αλλά δεν είμαστε και αισιόδοξοι για το πώς θα καταλήξει μια διαπραγμάτευση που ο κύριος παράγων η Βραζιλία δεν επιθυμεί επουδενή να ξεφύγει από την ελληνική που δείχνει με τις υπόλοιπες χώρες του Μερκοσούρ. Και αυτό που φαίνεται στις δικές μας τις σκέψεις και συζητήσεις και τις δυνατότητες μια συμφωνία με το Μερκοσούρ να γίνει μια διμερή συμφωνία με τη Βραζιλία νομίζω ότι μπορεί να ισχύσουν μετά από όσα υποστηρίζουν πολιτική κύκλη στη Βραζιλία, κυρίως ο Υπουργό Εξωτερικών. Λοιπόν, θα πρέπει να προχωρήσουμε το διάλογο στα πλαίσια του Μερκοσούρ, γνωρίζοντας όμως κάθε δυσκολία που αντιμετωπίζουμε, τις δυσκολίες με εκείνου αλλά και ανάμεσα σε εκείνου, γιατί μας ανησυχεί ιδιαίτερα και η θέση της Αργεντινής και ανησυχεί και τι αρχέ τη Βραζιλίας η στάση τη Αργεντινή. Όλα αυτά που σύντομα σας είπα θα μπορούσα να καταλήξω ότι υπάρχει ανάγκη εμείς ε, σαν Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και σαν Κοινοβούλιο να λάβουμε τις ευθύνες ε, μιας βαθύτερης ε, λεπτομερούς εξέτασης του θέματος αυτού και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι σε θέση να υιοθετήσει μια στάση συγκεκριμένη, οριστική πάνω σε αυτό που να είναι και η κατεύθυνση, ο προσανατολισμός, ο δημοκρατικός της Ευρώπης μας απέναντι στο Συμβούλιο και είναι περίπλοκοι οι παράγοντες οι εμπορικοί και οι πολιτικοί στο σύστημα αυτό σχέσεων και όπως γνωρίζουμε όλοι θα είναι μια τεράστια συμφωνία σύνδεση συνεργασίας που θα συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο πρόεδρος, ο τώρα. Uh, ε, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Σούστα για την ε, πολύ ενδιαφέρουσα ενημέρωσή του στο θέμα της παρακολούθησης εποπτικής ομάδας, ε, γιατί ακριβώς δείχνει ε, τη χρησιμότητα της εποπτικής ομάδας ε, σε σχέση με την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, γιατί έχουμε τη δυνατότητα, σε αυτή την εποπτική ομάδα μπορούμε να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες ορισμένων πτυχών. Κάτι ακόμη όμως θα ήθελα να πω, που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για μας, με την εμπειρία των διμερών ε, συμφωνιών ε, με, το, την Κολομβία και το Περού που είχε ως αποτέλεσμα ε, ο εταίρος μας ε, να είναι ένας περιφερειακός εταίρος σημαντικός, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε αν η Βραζιλία βγει από τη Μερκοσούρ, πρέπει να σκεφτούμε ότι το Μερκοσούρ είναι ένας περιφερειακός εταίρος, η προσέγγιση αυτή πρέπει να διατηρηθεί και Ο στόχος μας δεν πρέπει να είναι να επαναχωρήσουμε στην ιδέα της περιφερειακής συνεργασίας, αλλά να αναπτύξουμε περαιτέρω την περιφερειακή συνεργασία, γιατί έχουμε όφελος να λειτουργεί σωστά η Mercosur η οικονομική συνεργασία μεταξύ ε, των χωρών της Μερκοσούρ είναι υποφελής και για μας. Όταν μιλάμε για την Κίνα, μιλάμε για μια μεγάλη αγορά και έχει διαφορετικές ε, ε, τοπικές οντότητες με, διαφορετικές, με διαφορετικά συμφέροντα. Διαφορετική λοιπόν περίπτωση είναι η Κίνα και διαφορετική περίπτωση είναι η Μερκοσούρ. Γι' αυτό νομίζω ότι οι σχετικές ε, διαπραγματεύσεις και συνομιλίες πρέπει να προωθήσουν την περιφερειακή συνεργασία. Ευχαριστώ. Δεν είναι και τόσο αισιόδοξο άρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ούτε και στο Συμβούλιο ούτε και από το Μερκοσούρ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πάντα ε, ήταν ενθουσιώδης για το θέμα του Μερκοσούρ. Μήπως θα μπορούσε να μας δώσει, να μας προσφέρει μια ακτίδα φωτός και ελπίδας. Ούτε. Ναι, ναι, ναι, Δεν θέλω να σας τριμώξω. Πάνω σε αυτό ήταν ιδιαίτερα δραστήρια ενεργή η Επιτροπή Ευρωπαϊκή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, θέλετε ελπίδα. Όταν αναστούμε επίπεδα πάντα στρεφόμαστε προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα για την ερώτησή σου ότι έγινε προσφάτα ένας γύρο διαπραγματεύσεων για το Μερκοσούρ στην Βραζίλια. Είχαμε και μια αποπτική ομάδα σε επίπεδο κοινοβουλίου, στην οποία έδωσε η Επιτροπή πιο πολύ λεπτομερεί πληροφορίε. Βέβαια, οι διαπραγματεύσει με τη Μερκοσούρ είναι διμερεί σχέσεις από περιφέρεια προς περιφέρεια. Και επεσήμανε ο κύριος Σούλτς τις δυσκολίες που έχουμε σε επίπεδο εταίρων Μερκουσούρ στις διαπραγματεύσεις αυτές. Παρακολουθούμε λοιπόν εκ του συνεχείς διαπραγματεύσεις αυτές και θα ενημερώσουμε το Κοινοβούλιο για όποιες εξελίξεις λάβουν χώρα είναι προφανές νομίζω ότι καθώς η Μερκοσούρ είναι και αυτή η τελωνιακή ένωση, είναι μάλλον τελωνιακή ένωση, έχουμε δεσμούς που ξεπερνούν τις σχέσεις μας με άλλες περιφέρειες. Άρα θέματα που έχουμε με άλλες περιφέρειες δεν εφαρμόζονται απαραίτητα ε, αυτά καθεαυτά αυτά στις σχέσεις μας με την Μερκοσούρ. Ευχαριστώ πολύ. Προτείνω τώρα να ακούσουμε τον κύριο Σάλμπα, τον συνάδελφο για την επίσκεψη στην Κωνσταντίνα και τον Παναμά. Ναι. Μαζί με την αντιπροσωπεία για την Κεντρική Αμερική πήγα στον Παναμά και στην Κωνσταντίνα. Όλοι σας γνωρίζετε αυτή η συμφωνία σύνδεσης που την Ολομέλεια του Δεκεμβρίου θα ψηφιστεί και θα εγκριθεί, θα επικυρωθεί από όλα τα κοινοβούλια των χωρών της Κεντρικής Αμερικής. Προς το παρόν μόνο η Νικαράγουα έχει εγκρίνει, έχει επικυρώνει σε αυτή την ε, συμφωνία και σε σχέση με εμά. Για τον Παναμά είναι αρκετά αισιόδοξη η κατάσταση. Αντιθήκαμε με τον Υπουργό Εξωτερικών, με τον Υπουργό λοιπόν και μας διαβεβαίωσε ότι το Κοινοβούλιο του Παναμά θα επικυρώσει το Νοέμβριο μάλλον και τουλάχιστον όχι αργότερα, όχι μετά το Δεκέμβριο ώστε να μπορέσει και να ισχύσει προσωρινά και στον Παναμά και στην Καράγουα στα πλαίσια αυτά σε προσωρινή φάση τουλάχιστον ο Παναμάς επίσης είναι η μοναδική χώρα της Κεντρική Αμερική που δεν έχει αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή, της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης στην πρωτεύουσά του. Και με τα μέλη της κυβέρνησης της ζήτησαν μήπως θα μπορούσαμε να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ανοίξει μια αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκή Ένωση στον Παναμά μου προκάλεσε εντύπωση αυτή η κατάσταση. Είναι από τι χώρε με την περισσότερη δυναμική και με το ισχυρότερο ποσοστό ανάπτυξη στην περιοχή. Και θεωρούν ότι είναι κάπω αποκλεισμένοι γιατί δεν έχουμε εκεί εμεί αντιπροσωπεία. Αυτό λοιπόν θα μπορούσαμε να κάνουμε και θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Και μα είπε το Κοινοβούλιο ότι από οικονομική πλευρά θα μπορούσε να συνεισφέρει στην ε, στην αντιπροσωπεία αυτή που θα μπορούσε να ανοίξει στον Παναμά και επίσης ε, τι διαβεβαίωσή τους θα μπορούσε να επικυρώσει αυτά τα βήματα και ε, ταυτόχρονα ε, να δείξουμε το ενδιαφέρον μας για μια αντιπροσωπεία για την Κωνσταντίνα. Η κατάσταση όμως για την έγκριση της, για επικύρωση της συμφωνίας είναι κάπως περισσότερο περίπλοκο γιατί εκεί η κυβέρνηση δεν έχει καμία δυνατότητα πέρα από συγκεκριμένες στιγμές να επηρεάσει τα όσα σημαίνει στο κοινοβούλιο και τι σημαίνει αυτό. Τα πολιτικές ε, ομάδες της Κοσταρίκα είναι εκείνες που αποφασίζουν πότε θα προωθηθεί η επικύρωση της συμφωνίας. Ήταν σε επαφή με επιχειρηματικούς κύκλους, με τον κυβέρνηση, με την Υπουργό Εμπορίου και όλοι τους μας είπαν ότι είναι σημαντικό οι εθνικοί τους βουλευτές στην Κωνσταντίνα να τα διαπιστώσουν όλα αυτά ότι είναι ακριβώς πολύ σημαντικό να επικυρωθεί όσο γίνεται συντομότερα αυτό αυτή η συμφωνία ή μάλλον τα αρνητικά που θα έφερνε μια μη επικύρωση της συμφωνίας στην οικονομία της Κωνσταρίκας. Είναι μια προσωρινή έγκριση από τις χώρες που ήδη έχουν εγκρίνει και όσοι δεν το έχουν κάνει θα ε, έχουν αργότερα τη συμφωνία τα θετικά από όλα αυτά και υπάρχουν και ποσοστώσεις που δεν μπορούν να ισχύσουν από τώρα για αυτές τις χώρες αλλά οι υπόλοιπε χώρες που ήδη έχουν εγκρίνει θα μπορέσουν να υποφεληθούν από τις ποσοστώσεις τις δικές τους που δεν έχουν ακόμα επικυρώσει. Αυτά. Και μας είχαν πει ότι η έγκριση, θα, η επικύρωση θα γινόταν ε, στην αρχή τουλάχιστον 2013, αλλά αυτό θα ήταν αρνητικό για τα οικονομικά συμφέροντα της Κωνσταντίνα. Και οι βουλευτές πάντως έδειξαν ότι είχαν διάθεση να επικυρωθεί η συμφωνία αυτή το πρώτο τρίμηνο του 2013. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό, θετικό σημείο. Και ακόμη κάτι μαζί ζήτησε η κυβέρνηση Κωνσταντίνα να τους βοηθήσουμε για την υποψηφιότητά τους στον ΟΣΑ. Η Κολομβία και η Κοστορίκα είναι υποψήφια μέλη για την οικονομική συνεργασία και ανάπτυξη και φαίνεται ότι για γεωπολιτικούς λόγους οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν μόνο την Κολομβία και εκείνοι μας είπαν μήπως θα μπορούσατε εσείς να υποστηρίξετε την είσοδο και της Κοσταρίκα. Έτσι. Και θα θέλαμε λοιπόν αν συμμετάσχουμε θα ήταν κάτι το ιδιαίτερα θετικό για αυτούς. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτά ήθελα να πω. Κάποια ερώτηση παρακαλώ. Κάποιο σχόλιο από πλευρά τη Επιτροπή. Όχι, το επόμενο σημείο. Ο Λάγκε είναι σχεδόν ο μόνος από εκείνου που πήγαν ε, από το κοινοβούλιο στη Ρωσία και μόλι ξέφυγε από τους ατμούς Βότκα που εισέπνευσε <laughs> λοιπόν για πέστε μα τι αποκομίσατε σαν ε, <laughs> εντυπώσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έρευσε πολύ βότκα. Είχαμε πολύ πυκνό πρόγραμμα από τη γραμματεία οργανωμένο. Συναντηθήκαμε με εταίρους από κάθε επίπεδο, από την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία, τη Ρωσική Βιομηχανία, βουλευτές της Ντούμα, Συζητήσαμε με εκπροσώπους Τελωνιακής Ένωσης, με την Λευκορωσία και το Καζακστάν, εκπροσώπους της κυβέρνησης. Επομένω είδαμε σε κάθε επίπεδο φορείς και παράγοντες της ρωσικής ε, πλευράς. Βεβαίως πάνω απ' όλα συζητήθηκε το θέμα της προσχώρησης της Ρωσίας στο ΠΟΕ. Βεβαίως και είχαμε θέματα των εφισταμένων ακόμη εμπορικών εμποδίων, εμπορικών φραγμών και θέματα της ενεργειακής συνεργασίας. Εάν θέλετε να σας πω τι βλέπω στο πηλίκον, πρέπει να πω ότι η στάση της ε, ε ρωσικής πλευράς απέναντί μας ήταν μάλλον λόγος απότομου ξυπνήματος θα έλεγα, γιατί και λόγω της των οικονομικών μεγεθών της ε, ρωσικής ε, πλευράς ε, θεωρούν ότι μπορούν να συμπεριφερθούν όπως θεωρούν εκείνοι σκόπιμο. Βλέπουμε ένα power play όπως ονομάζεται, δηλαδή μια διελκυστίνδα δυνάμεων. Έχουμε επί παραδείγματι τον Υπουργό, ο οποίο μα είπε ότι εάν θέλουμε να είμαστε εταίροι, πρέπει να συμπεριφερόμαστε και σαν εταίροι απέναντί του και μας ε, μίλησε για το θέμα του αγωγού Ναμπούκο κατά τρόπον αρκετά πιεστικό. Πρέπει να πω ότι ήταν ένα απότομο ξύπνημα για μένα αυτό και δεδομένης και της γεωπολιτικής κατάστασης, μια και συστήσαμε μόλις τώρα το θέμα της ε, Κίνας, δεν βλέπω πολλές ελπίδες να γεννιούνται από την ε, τελευταία αυτή επαφή με την Ρωσία. Δεν μπορώ να στηρίξω πολλές ελπίδες σχέση με τη Ρωσία και επίσης σε θέματα που έθιξαν οι εταίροι για το τρίτο πακέτο για την ιστορική αγορά, την, ενέργεια, την ιστορική αγορά της ενέργειας ή το θέμα της νομοθεσίας για την ε, χημεία, για τα χημικά προϊόντα. Ε, είδαμε πολλές αντιδράσεις και από πλευράς Ρώσων πολλούς περιορισμούς που επιβάλλονται. περιορισμούς οι οποίοι στόχο έχουν να αντισταθμίσουν απώλειες ε, που προκύπτουν ενδεχομένω από την προσχώρηση των ΠΟΕ και την μείωση των τελωνιακών δασμών. Φερρυπίν, εισάγεται ένας φόρος ανακύκλωσης για τα ιδιωτικά ιδιωτικής αυτοκίνητα μόνο όμως τα εισαγωγής, όχι στην τοπική παραγωγή. Είναι προφανές ότι αυτή η ειδική νομοθεσία αυτή, η ειδική φορολογία επιβάλλεται προκειμένου να ε, ενισχυθεί η εσωτερική, παραγωγή και να εμποδιστούν οι, οι εισαγωγέ ή να γίνουν πιο ακριβέ. Επομένω βλέπουμε μια τέτοια συμπεριφορά από πλευρά, ε, Ρώσων, την οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη και αναλόγω να τη δράσουμε. Ευχαριστώ. Νομίζω και ο κύριος Δαβίδ ήταν μέρος της αντιπροσωπείας αυτής. Θέλετε να πείτε κάτι. Ευχαρι... Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω να πω τίποτα. Απλώ ότι είδαμε το πρώτο χιόνι τη χρονιά. Το πρώτο χιόνι για φέτο. Μάλιστα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Merci. Nous passons au point 8 euh, et 9. Περνάμε στο σημείο 7. Au niveau du draft Euh, euh, Όσον αφορά τις ε, πτυχές ε, της ανάπτυξης, ε, για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε θέματα γενετικών πόρων και ειδικότερα τις επιπτώσεις στη μείωση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Χέλμουντ Σόλτσο, η συζήτή μας. Είναι θέμα πολύ σημαντικό και για τη δική μας Επιτροπή αλλά και για την Επιτροπή Ανάπτυξης ε, που είναι ο καταμερισμός του ωφέλους ε, από τους γενετικούς πόρους. Προτείνω λοιπόν ο Χέλμου να μας πει ορισμένα πράγματα για το πώς έχει η κατάσταση το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής είχαμε μια διεξοδική συζήτηση ως προς τις γενικές πτυχές του θέματος. Γνωρίζουμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολλές επιτροπές, όχι μόνο την Επιτροπή του Εθνικού ή την Επιτροπή Ανάπτυξη που συζητήθηκε. Αλλά έχουμε να κάνουμε πτυχέ ε, των εμπορικών συναλλαγών και τις σχετικές συνέπειες. Έχουμε λοιπόν για την Επιτροπή Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της ε, προσπαθήσει να προβάλλουμε αυτές τις πτυχές σημειώνοντας ότι είναι πολλές οι πτυχέ τις οποίες ακόμη θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε στη γνωμοδότηση αυτή και ξέρω ότι όλοι οι συνάδελφοι γνωρίζουν ότι κατά την κατάθεση μιας, προτάθεσης, μιας προτάσεως γνωμοδότησης είμαστε υποχρεωμένοι να περιοριστούμε μόνο σε ορισμένες ε, θέσεις, δεν μπορούμε να περιλάβουμε τα πάντα. Πάντως θέλω να πω ότι με πολύ ενδιαφέρον περιμένω να συναντήσω τους σκιώδεις ηγητές για να προβούμε σε μια εντατική συνεργασία ως προς το τι μπορούμε να περιλάβουμε σε στην γνωμοδότηση ώστε αυτή να εμπλουτιστεί προς την κατεύθυνση που θεωρούμε ε, σκοπιμότερη και καταλληλότερη. Και θα θέλω να αναφερθώ συμπληρωματικά σε σχέση με τις συνεδρίες του Οκτωβρίου στις εξής πτυχές γιατί έχουμε να κάνουμε ουσιαστικά με το πώς θέλουμε τις, ε, τα έσοδα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό στην την TRIPS, ε, τον ΠΟΕ, να τα χειριστούμε και πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε τις ιδέες αυτές στην γνωμοδότηση της Επιτροπής ε, Ανάπτυξης. Επίσης, η γύρι ε, συνεννόησης, συνδιαμόρφωσης ε, συντονισμού και τις διαπραγματεύσει θα πρέπει πιστεύω να οργανωθούν κατά τρόπο και νομικά βέβαια ορθό αλλά και ε, ικανό να επηρεάσουν ουσιαστικά τις διαπραγματεύσεις αυτές και να έχουμε μια κατάσταση τόσο νομικά στέρεα όσο και διαφανή. Επίσης, δεύτερο σημείο, θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα του PIC, των ε, αρχών δηλαδή των, ε, της συνένεσης μετά από ενημέρωση, που ήδη βλέπουμε στο πρωτόκολλο της Ναγκόια, δηλαδή ότι υπάρχει μια θέση διεθνώς νομολογημένη, αλλά την οποία δεν έχουν ε, τα κράτη-μέλη στην ουσία υλοποίηση. Δηλαδή, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει και δεσμεύεται για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου στην Αγκόγια, αυτή η δέσμευση είναι και υποχρέωση για τα κράτη-μέλη να το εφαρμόσουν. Και νομίζω και στην περαιτέρω επεξεργασία του θέματος θα πρέπει να μιλήσουμε μόνο ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο αλλά και τα κράτη-μέλη επιμέρους είναι δεσμευμένα να προχωρήσουν σε μια ταχεία ε, κύρωση του, της σχετικής νομοθεσίας, του πρωτοκόλλου δηλαδή της Ναγκόια. Τρίτον, συνεχίζονται βεβαίως οι συνομιλίες, συνεννοήσεις κτλ ιδιαίτερα στο πλαίσιο όσον αφορά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματική Διοκτησία. Και νομίζω ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη ε, συντονισμένα, ύστερα από συνεννόηση, να τοποθετούνται και να υπογραμμίζουν ότι πρέπει μια υπουργική ε, διάσκεψη του ε, ΠΟΠΗ να δώσει τις θέσεις ε, να συζητήσει και να καταλήξει σε αποφάσεις τα θέματα που μας απασχολούν. Και τέταρτον, το ζήτημα της αηφόρου ανάπτυξης στα τρίτα κράτη και η θέση η δική μας σε σχέση με τους αυτόχθονες ε, λαούς και την κατάσταση προκύπτει μετά τις νέες Εθνής ε, συμφωνίες. Άρα λοιπόν θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να προσφέρουμε μια προοπτική για την επιβίωση των αυτοχθόνων λαών. Αυτό είναι νομίζω μια άλλη πτυχή της ανάπτυξης και των ε, εμπορικών ε, σχέσεων που θα πρέπει να συζητηθεί και να προβληθεί. Αυτό το καταγράφω εν συντομία στο σημείο 5, προσπαθώντας να είμαστε δυνατόν πιο σύντομος. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη συνεργασία. Έχουμε πολύ στενά χρονικά όρια και ελπίζω παρ' όλα αυτά ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια καλή πρόταση ώστε στη δεύτερη σύνοδο του Νοεμβρίου να μπορέσουμε να εγκρίνουμε το κείμενο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος για την τροπολογία προθεσμία 8 Νοεμβρίου στις 6. Σκιώδης εισηγητός. Κρίστοφερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν έχω και πολλά να πω γιατί νομίζω ότι είναι πολύ καλό το ε, σχέδιο ε, γνωμοδότησης νομίζω ότι είναι πολύ εξισορροπημένο. Θέλουμε κάπως να το περιορίσουμε, όπως είπε και ο Χέλμουτ, στις ε, ε, πτυχές που αφορούν ειδικότερα την Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορίου. Ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις, τροπολογίες από πλευράς Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι αυτό το κείμενο που έχουμε μπροστά μας περιλαμβάνει τις βασικές γραμμές που θα ακολουθήσουμε. Ε, είναι πραγματικά ειλικρινές στο σχολείο μου όταν σας λέω ότι έχετε την υποστήριξή μου και είναι σπάνιο εκ μέρους μου. Εντάξει, πολύ καλά. Σόλν και Φέλνερν, ναι, πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα πρέπει να εγγραφεί στα πρακτικά και να το επικυρώσουν οι πολιτικές ομάδες για την επόμενη συνάντηση. σοσιαλιστές. Ο συνάδελφος, η συνάδελφος, συγγνώμη. Ναι, να συγχαρώ. Πρόκειται για ένα θέμα με προβλήματα όμως, ενδιαφέρει και άλλες επιτροπές. Εμείς θα πρέπει να δούμε την εμπορική πτυχή και είναι γνωμοδότηση. Θα πρέπει να δούμε το εύρος του κειμένου. Ορισμένες αποχρώσεις όμως και ορισμένα στοιχεία που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε για να δούμε τι ζητάμε απέναντι σε αυτή την πνευματική διεκτησία, τη Διεθνή Συμφωνία και τον ορισμό τι σημαίνει πειρατεία αυτών. Ε, θα πρέπει να δούμε αυτά ξεκινώντας για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται για να δούμε αυτός ο κόσμος πώς θα ωφεληθεί, είναι αναπτυσσόμενος ε, από τις εμπορικές σχέσεις ε, και από όλα αυτά που να συμμετέχουν όλοι στη συμφωνία και για τη βιοπικιλότητα και καινοτόμες λύσεις ε, να ε, πέρα από τις άδειες εκμετάλλευσης επειδή όλα αυτά σημαίνουν τεχνικές δυσκολίες ε, για τις συμφωνίες ανάμεσα στις χώρες προέλευσης και τις χώρες που θα υποφεληθούν και πρέπει να μιλήσουμε για εμπόριο σπόρας, σπόρων. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχουν ορισμένοι που έχουν ειδικέ άδειε εκμετάλλευση και να πρέπει να δούμε τα εξή πράγματα. Τη βιοπικιλότητα, εξασφάλιση διατροφής και δυνατότητα ε, ενός εμπορίου για τους γεωργούς που ασχολούνται με τις νέους σπόρους. Ε, νομίζω ότι συμφωνείτε ότι είναι κάπως περισμένο το κείμενο και με κατάλληλες ε, τροπολογίες θα του δώσουμε τα κατάλληλα χρώματα για να βελτιωθεί. Διαφορετικά θα είναι αρκετά καλό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Φραντσίσκα Κέλλερ για τους πράσινους. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι σκιώδης συγγήτρια. Η Εμίλια είναι, αλλά δεν μπορεί να είναι εδώ δυστυχώ. Σε γενικές γραμμές και οι πράσινοι υποστηρίζουν ε, την γνωμοδότησή σου, Χέλμουτ. Πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ καλή βάση συζήτησης Απλώ πιστεύουμε ότι κάποια ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά παραμένουν ανεπίλητα στη γνωμοδότηση αυτή, αλλά δεν ξέρω, ίσως ενδεχομένω ε, η Επιτροπή ανάπτυξη ε, να έχει ασχοληθεί περισσότερο με αυτό, το κατά πόσο η γενετική πόρη θα έπρεπε να είναι αντικείμενο ευαισθητεχνίας ή όχι και αν ναι, ε, σε τι επίπεδο εφαρμογών, Πώ μπορούμε να δώσουμε μια αποτελεσματική φωνή στα συμφέροντα των τοπικών κοινοτήτων. Οι γυναίκε, για παράδειγμα, είναι μεταξύ των ενεργών χρηστών ε, γενετικών πόρων ε, για λόγους αναπαραγωγικής υγείας, πώς μπορούμε λοιπόν να ε, εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή τους, πώς ορίζουμε την παραδοσιακή γνώση. Και αυτό είναι ένα ερώτημα αφετηρία. και πώς ε, δεν, ε, δεν δημιουργούμε ένα βάρος ε, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ένα ιδιαίτερο κόστος για τις αναπτυσσόμενες χώρες και μιλάω ειδικότερα για τις συμφωνίες TRIPS. Όλα αυτά τα ζητήματα πιστεύουμε ότι μπορούν να απαντώνται στο πλαίσιο μιας τέτοιας γνωμοδότησης. Ενδεχομένω η Εμίλια να υποβάλει κάποιε τροπολογίε προ αυτή την κατεύθυνση, αλλά σε γενικέ γραμμέ είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την έκθεσή σα. Ευχαριστώ η Κατρίν. Η Κάθριν. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να προσθέσω τη δική μου υποστήριξη στην ε, έκθεση αυτή. Άλλωστε πολλά από όσα ήθελα να πω έχουν ήδη υποθεί. πρέπει να έχουμε μια προληπτική προσέγγιση όταν έχουμε να κάνουμε με, τους, ε, με τις ε, γενετικές ε, τροποποιήσεις και σκέφτομαι ιδιαίτερα με την επιβολή, αν έχουμε κανόνες δηλαδή, πώς θα επιβάλλονται. Αυτό με απασχολεί ιδιαίτερα. Αλλά η έκθεση αυτή είναι πραγματικά, έχει πραγματικά μία πολύ ε, σωστή και εξισορροπημένη προσέγγιση και θα έπρεπε να ευχαριστήσουμε τον εισήγητη γι' αυτό. Υπάρχει βέβαια πάντοτε το κόστος ε, της έρευνας ε, και της εφαρμογής της και των ανοιχτών πηγών και όλα αυτά σε σχέση με την βιοπικιλότητα. Ε, αυτό το θέμα παραμένει. Το λέμε κυρίως για την κυκλοφορία των προϊόντων που έχουν τροποποιηθεί γενετικά και όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να μας απασχολούν. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ενδεχομένως λοιπόν υποβάλλουμε κάποιες τροπολογίες σχετικά, αλλά δεν θα είναι πολλές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Από πλευράς Επιτροπής... Διακόπτει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, έχουμε και εκπροσώπους από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Ο κ. Κουτσούρης ή Μπέκ, κάποιος από τους δύο θα επιθυμούσε το λόγο. Thank you. Um, uh, Ευχαριστώ και καλημέρα σας. Λίγες παρατηρήσεις μόνο. Πιστεύουμε ότι είναι μια ισορροπημένη πρόταση γνωμοδότησης. Ένα πράγμα θα ήθελα να υπογραμμίσω, που ίσως θα ήταν καλό να εξεταστεί. Εξετάζουμε τη γενική μας διεύθυνση το θέμα των γενετικών πόρων πολύ ευρύτερα, όχι μόνο από την έποψη των πνευματικών δικαιωμάτων. Κοιτάμε λοιπόν τη γενικότερη εικόνα και όχι μόνο το ένα θέμα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και όλες οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έχουν συναντηλήψει ότι έχουμε να κάνουμε με θέματα κοινού συμφέροντος όλων των κρατών, όλων των ερευνητών ώστε να έχουμε ένα σύστημα ανοιχτό, ένα σύστημα που θα επιτρέπει την ανταλλαγή και χρήση γενετικών πόρων και τις συναφούς παραδοσιακής γνώσης που αποτελούν βάση για έρευνα, καινοτομία βασισμένη στην ε, βιοπικιλότητα και τους γενετικούς πόρους. Βεβαίως αυτό με σεβασμό των δικαιωμάτων εθνική κυριαρχία των κρατών, αλλά και των δικαιωμάτων των ηθαγενών πληθυσμών. Το δικαίωμα δηλαδή στην παραδοσιακή γνώση. Πάντως είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι το θέμα δεν αφορά σχέσεις μόνο βορρά-νότου. Δεν πρόκειται για μια αντιπαράθεση ως προς την ανάπτυξη μόνο. Έχει μια εγκάρσια παρουσία και σημασία. Ένα παράδειγμα. χώρες του, για τις χώρες του ΩΣΑ θεωρείται ότι μπορεί να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το γενετικό υλικό για την ε, γεωργία. Και όμως ο λόγος είναι αντίστροφος ότι οι κύρια εξαρτώμενες χώρες είναι οι χώρες του Νότου που εξαρτάται από τους γενετικούς σπόρους των βορείων κρατών, κυρίως όσον αφορά τους γενετικούς σπόρους του ζωικού κεφαλαίου. Αυτό που θέλω δηλαδή να εξηγήσω είναι ότι δεν πρόκειται για μια καθαρή αντιπαράθεση μεταξύ βορρά-νότου. Υπάρχουν βεβαίως πτυχές βορρά-νότου, αλλά ένα ζήτημα εγκάρσιο, ένα ζήτημα όπου όλες οι χώρες έχουν κοινό συμφέρον να βρουν ε, ένα πλαίσιο που θα τους επιτρέπει να λειτουργούν και να δρούν. Για δε την κύρωση του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια που έφυγε νωρίτερα. Θα θυμάστε, ίσως θα γνωρίζετε, πως υπάρχει μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ευρωπαϊκό κανονισμό εφαρμοστικό στο πρωτόκολλο Ναγκόγια που θα μπει τώρα κατά την άποψη της Επιτροπής στην τακτική νομοθετική διαδικασία, στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δηλαδή θα υποβληθεί. Αυτή η τακτική διαδικασία είναι για μας προϋπόθεση για να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη στην κύρωση του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια. Ευελπιστούμε δε ότι είναι δυνατόν να επιταχυνθεί ε, και να προχωρήσει προσκόπτα μια τέτοια νομοθετική διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ ο Χέλμουτ για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ σύντομα. Ευχαριστώ σύντομα. Ευχαριστώ για όλα τα σχόλια. Με την ε, τοποθέτηση Επιτροπής σήμερα, πιστεύω, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πιστεύω μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις ε, λεπτομέρειες για την προσεχή της Επιτροπής μας, ώστε να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε την ψηφοφορία. Καταγράφω τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν και θέλω να υπογραμμίσω για μια φορά ότι από τη δική μου άποψη σημασία έχει να ανοίξουμε το οπτικό μας πεδίο και να κοιτάμε τα γενικότερα ζητήματα. Βεβαίω αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν προσδοκίες, ελπίδες και το καθεξής για να αντιμετωπίσουμε αυτό το σημαντικό και δύσκολο ίσως θέμα, αλλά πρέπει και να επικεντρωθούμε στα πραγματικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις, που σχετίζονται με αυτές τις διεθνείς ε, δεσμευτικά και δεσμευτικές συμφωνίες. Και ως εκ τούτου πρέπει και να εμπλουτίσουμε αντίστοιχα την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης, την οποία δεν αμφισβητώ, διότι θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ καλές πτυχές ήδη, νομίζω ότι θα πρέπει να συμπληρώσουμε κάποια δικά μας θέματα την πρόταση αυτή και ιδιαίτερω δεν θέλω να ευχαριστώ την κυρία Ρόντεμπεκ, την Μύρια της Γραμματείας, διότι ιδιαίτερα, ιδιαίτερα μας βοήθησε στην διατύπωση του κειμένου. και μας επιτρέπει με τη βοήθειά της να ευελπιστούμε για καλά αποτελέσματα στην προσοχή συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. κάνει, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για το θέμα αυτό. Οκτώ και 9 εμπορική κοινωνική ευθύνη δύο θέματα. 25 Οκτωβρίου 2011 υιοθέτησε μια ανακοίνωση Επιτροπή για τη νέα στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση 2011-2014 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και το Κοινοβούλιο ανταποκρίθηκε ιδιαίτερα. Η Επιτροπή μας, η Απασχόλησης και η Νομική Επιτροπή ε, ανέλαβαν εκθέσεις πρωτοβουλίας. Ο καθένας ε, έχει βέβαια και δικαίωμα έκφραση άποψη για την έκθεση του άλλου. Έτσι μπορούμε να επεξεργαστούμε ιδιαίτερα και κατάλληλα το θέμα. Ο Ντεζίρο, ο οποίος ε, τους εκπροσώπους και στον Μπερτ Λάγκε έδωσε αυτή την έκθεση γνωμοδότησης, ε, τη μεταβίβασε φεύγοντας, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι το Όντι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στην ανακοίνωση, κατέθεσε την ανακοίνωση που μας περιέγραψε ο Πρόεδρος, η οποία δείχνει μια αλλαγή στρατηγικής για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, η οποία μέχρι τώρα ήταν ε, επικεντρωμένη λίγο πολύ σε μια εκούσια συμμετοχή, σε θελοντική συμμετοχή. Τώρα βλέπουμε πιο ε, δεσμευτικούς όρους στην, ε, στις προϋποθέσεις ε, και στην αντιμετώπιση του θέματος εταιρική κοινωνική ευθύνη. Με δύο παραδείγματα. Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε παραδείγματι, καλούνται τα κράτη-μέλη στα τέλη του 2012, δηλαδή πολύ λίγος καιρός ακόμα μένει, να καταθέσουν για τις εθνικές τους επιχειρήσεις προγράμματα για την ε, κοινωνική εταιρική, ε, εταιρική κοινωνική ευθύνη, τα οποία θα επεξεργαστούν από κοινού με, την, με τις επιχειρήσεις με των επιχειρήσεων. Επίσης, μέχρι το 2015 προβλέπεται στην ανακύρωση της Ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ισχύουν τέτοιου είδους δεσμευτικοί όροι για όλες τις επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να έχει γίνει προσαρμογή στο διεθνές πρότυπο ISO 26.000 ή στα διεθνή πρότυπα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια εξέλιξη και πλέον δεν είναι ε, κούσια ε, και κατατοδοκούν η ανάληψη εταιρική κοινωνική ευθύνη για τι επιχειρήσει μα. Και γιατί. Διότι, αγαπητοί συναδέλφοι, αν δούμε πώ οι επιχειρήσεις μας συμπεριφέρονται σε κάποια κράτη του πλανήτη, τότε δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι δεν ακολουθούν, δεν τηρούν προδιαγραφές και όρους που ισχύουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρόκειται για την Αφρική, δεν πρόκειται για την Ασία, δεν πρόκειται για τη Ρωσία ακόμη. Βλέπουμε ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, πολύ συχνά παραγνωρίζουν όσο μπορούν την νομοθεσία για τα κοινωνικά, για τα εργασιακά και επομένως, ε, δεδομένου ότι και εμείς θέλουμε να ε, ακολουθήσουν τα άλλα κράτη εταίροι, τα άλλα κράτη του κόσμου, τι προδιαγραφέ των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή του ε, Διεθνού Οργάνου εργασία για τα εργασιακά, το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα είναι να απαιτούμε από τι ευρωπαϊκέ μα επιχειρήσει όταν δραστηριοποιούνται έναν τον κόσμο να τηρούν τι ίδιε αυτέ προδιαγραφέ. Και γι' αυτό υποστηρίζω την προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητώ στην έκθεση που σας έχω καταθέσει, να προχωρήσουμε λίγο ακόμα και αυτό γιατί καταρχάς πιστεύω ότι μια εμπορική ε, συμφωνία διεθνής στο μέλλον θα πρέπει ιδιαίτερα να υπογραμμίζει αυτές τις αρχές ε, της εταιρείε κοινωνική ευθύνη για τις επιχειρήσεις μας, ε, στο πλαίσιο ιδιαίτερα της GSP και τη GSP+, των του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων και αντίστοιχα να προσαρμόζονται σε αυτές τις αρχές επιχειρήσει μα. μας. Επίσης, όταν βλέπουμε ότι η συμπεριφορά και η στάση των ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ανά τον κόσμο αμφισβητείται τόσο πολύ και ρητά από πολλές πλευρές θα πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα της δικαιοδοσίας, δηλαδή να είναι δυνατό να προσφύγει κανείς στα δικαστήρια, τα ευρωπαϊκά, για συμπεριφορά των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην διεθνή σκηνή. Και Τρίτον, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί μέχρι το 2014 όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να έχουν ε, ευθυγραμμιστεί στις προδιαγραφές περί εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, το 26.000 του ΙΖΟ ή το Global Contract συγκεκριμένα, τότε νομίζω ότι αυτονόητο είναι η προσαρμογή αυτή, η ευθυγράμμιση αυτή να γίνεται κατά τρόπο διαφανή. Και έτσι η υποχρέωση λόγοδοσίας στο πλαίσιο των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών αλλά και των ανωνύμων εταιριών θα πρέπει να ακολουθεί όχι μόνο, να καταγράφει όχι μόνο τις οικονομικές δραστηριότητες αλλά και την ε, εταιρική κοινωνική ευθύνη και να, κοινοποιείται, να τα σχετικά στοιχεία έτσι ώστε ο κάθε μέτοχος αλλά και ο κάθε πολίτης να είναι σε θέση να παρακολουθεί την συμπεριφορά της εν λόγω επιχείρησης. Και γι' αυτό Χαίρομαι ιδιαίτερω και περιμένω να ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων για το θέμα αυτό και βεβαίως αν έχετε κάτι να προσθέσετε στην πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Σκιώδη εισηγητέ. Φρασίσκα Κέλλερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μπέντ. Για την πολύ καλή σου πρόταση. συμφωνούμε απολύτω εμεί οι πράσινοι για τις ρήτρε εταιρική κοινωνική ευθύνης, δηλαδή στη διαπίστωση ότι δεν επαρκεί το να είναι κούσια η συμμόρφωση, πρέπει να είναι δεσμευτικέ, δεν μας αρκούν τα ωραία λόγια. Και πρέπει βεβαίως να εισαχθεί αυτή η, η έννοια και στα στις συμφωνίες ε, γενικευμένων προτιμήσεων και στην, ε, στις γενικευμένες προτιμήσεις plus, συν. Νομίζω ότι θα μπορούσε η Επιτροπή μας άλλωστε πολύ περισσότερο να συμβάλλει με μια καλύτερη συνοχή και συνέπεια ως προς το ζήτημα αυτό. Γιατί παραδείγμα τις οδηγίες για, την, ε, για τα λογιστικά ε, υπήρξαν κάποιες τροπολογίες που δεν πέρασαν, που αν είχαν εγκριθεί θα είχαν βελτιώσει σημαντικά ε, την νομοθεσία μας ως προς το θέμα της εταιρικής, ε, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Εν πάση περιπτώσει, πέρασε αυτό τώρα. Οι προτάσει του Μπέρντ Λάγκ μα ικανοποιούν. Έχουμε και εμεί του ίδιου του προσανατολισμού. Συμφωνίε δηλαδή με τρίτα κράτη πρέπει να είναι δεσμευτικές, να έχουν μια δεσμευτική ρήτρα ως προς την ε, τήρηση των κατευθυντηριών γραμμών των εθνών, πράγμα το οποίο επίσης θα σήμαινε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα κράτη εταίροι δεσμεύονται να εφαρμόζουν τις ε, κατευθυντήριες γραμμές. Επίσης κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε στην έκθεση θα ήταν ε, να αναθεωρηθούν οι ε, φυστάμενες ήδη συμφωνίες ώστε να ενσωματωθούν ρήτρε περί εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Οι δε ανά τον κόσμο πρεσβείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξέρουμε ότι έχουν εμπορικό ακόλουθο, ο οποίος ασχολείται με τις εμπορικές σχέσεις κτλ. Αλλά θα έπρεπε να έχουν, πιστεύουμε, και κάποιον ο οποίος ε, θα είναι ειδικευμένο, κατηρτισμένος ως προς το ε, ΕΚΕ, δηλαδή την εταιρική κοινωνική ευθύνη και να παρακολουθεί την εξέλιξη αυτών των ε, συμφωνιών, των διεθνών συμφωνιών και την τήρηση των όρων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Το ίδιο μπορεί να γίνει και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερική Δράσης, Ευρωπαϊκής Αρχής Εξωτερικής Δράσης. Ίσως θα μπορούσαμε να μεριμνήσουμε και για την καλύτερη εποπτεία της στηρίσης της ρήτας αυτής. Όπως είπες εσύ μιλάς για διαφάνεια. Εμείς λέμε ότι θα μπορούσαμε να, υπάρ... θα μπορούσαμε να και μια έννοια εποπτείας, να παρακολουθούμε ε, και να καταγράφουμε το κατά πόσον ε, εφαρμόζονται ε, οι διατάξεις. Ναι, κάποιες λοιπόν τροπολογίες, λίγες τροπολογίες, αλλά πάντως προς, τον ίδιο, προς την ίδια κατεύθυνση με σένα, Μπέρντ, και κυρίως για να ενισχύσουμε το κείμενο. Ευχαριστώ, η Κατρίν θα ήθελα να μας λάβει στο λόγο. Κατρίν, όχι. Ο Χέλμουντ τότε. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την ε, ε, πρόταση εκθέσεως. Ε, ο Πολ Μέρφυ είναι εκ μέρου μα, αλλά χρειάστηκε να πάει σε μια, ε, σκιώδη εισηγητής, αλλά χρειάστηκε να πάει σε μια άλλη συνεδρίαση αυτή τη στιγμή. Πάντω είναι πολύ σημαντικό το θέμα, Μα ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Στο σημείο 1, το οποίο βλέπω να έχει διατυπωθεί κατά πολύ ικανοποιητικό τρόπο, ε, ίσως θα έπρεπε να συζητήσουμε ιδιαίτερως πόσο είμαστε εμείς αρμόδιοι να συζητήσουμε τις συνέπειες της αγωγής των αρχών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Έχουμε και άλλη συναρμόδια επιτροπή πιστεύω, αλλά πρέπει να συστήσουμε και με την ΟΣΑ και με τα Ηνωμένα Έθνη. Πρέπει να δούμε δηλαδή σε διεθνέ επίπεδο, γιατί ναι, είναι κάπω αόριστη η διαμόρφωση, η διατύπωση των αρχών τη ΕΚΕ, αλλά στον ΟΣΑ ιδιαίτερω έχουμε περισσότερο δεσμευτικά κριτήρια, πιο σαφή κριτήρια και ίσω θα πρέπει να προσανατολίσουμε τι διαπραγματεύσει μα εμπορικέ ε, προ την κατεύθυνση αυτή για να δούμε αν μπορούμε να βρούμε κάτι πιο απτό σε επίπεδο ΟΣΑ που να αξιοποιήσουμε και για να προχωρήσω στη δεύτερη παρατήρηση, στο σημείο 6, Μπέρντ, ε, βρίσκω πολύ εύστοχη την ε, διατύπωση στην οδηγία περί διαφανείας. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να εισαγάγουμε επαρκή ΕΚΕ. Πολύ σωστά το λες. Δεν έδειξε αρκετή πυγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή τσαγανό ώστε να επιβάλλει αυτές τις ε, αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αλλά νομίζω ότι πέραν του να εκφράζουμε τη λύπη μας θα έπρεπε να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα και να πούμε τι άλλο μπορούμε ή θέλουμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Άρα θα έλεγα ότι θα, βά... θα... Εγώ πρότεινα να βάλουμε και ένα διατάφτα στην, ε, στην ε, παράγραφα 6. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Άντσλικ. Ευχαριστώ πρόεδρε κυρίες και κύριοι. Συγγνώμη για την καθυστέρησή μου, η κυρία Χάντσλικ. Αλλά μόλις τελειώσαμε στην Επιτροπή ΕΝΚΟ τις ψηφοφορίες. Μόλις ήρθα λοιπόν τώρα και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συντάκτη για όσα μας λέει και αυτές οι προϋποθέσεις είναι απαραίτητες που προτείνει ώστε η πολιτική αυτή να χαρακτηρίζεται από συνοχή σχετικά και με τους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τις αρχές του εμπορίου δεν θα πρέπει να διαφέρουν από άλλες προϋποθέσεις και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δημιουργήσουν υπερβολές όσον αφορά τις θεμελιώδεις ελευθερίας η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και του εμπορίου θα πρέπει αυτά στενά να συνδέονται μεταξύ τους. Υπάρχουν και συμφωνίες μεταξύ των κρατών και η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων βασίζεται όμως σε μια θελοντική βάση. Η σχέση μεταξύ των δύο, του εμπορίου και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων θα αποτελούσε σημαντικό βήμα για την ε, καλύτερη εφαρμογή αυτών των αρχών και οι επιχειρήσεις ακριβώς να μπορούν να σεβαστούν καλύτερα τα πρότυπα, τα κοινωνικά και τα παραβαλλοντικά και μέσω των κρατών. Το σύστημα αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδι για το διεθνές εμπόριο. Και όσον αφορά την Κίνα, Εκεί επίσης υπάρχει διάθεση σεβασμού αυτών των αρχών, αλλά χρειάζονται νομικές ε, αρχές. Ε, μια προσέγγιση στο σύστημα αυτό κατάλληλη ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να εφαρμόσουν αυτές τις αρχές και να τις στηρίσουν. Εδώ λέμε ότι θα πρέπει να αλλάξουν και τον τρόπο Ενεργεια τους, δράσεις τους ε, και για να σεβαστούν τα κοινωνικά πρότυπα, κυρίως σε τρίτες χώρες. Εμείς χρειάζεται ιδιαίτερα να τονίσουμε την πτυχή αυτή. Θα πρέπει να δούμε και την το μη σεβασμό αυτών των αρχών ότι αποβαίνει εις βάρος και των εργαζομένων στην Ευρώπη. Θα πρέπει να απαιτηθεί οι κοινωνικοί και οι περιβαλλοντικοί κανόνες να γίνονται σεβαστοί. Υπάρχουν πάντως δυνατότητες νέας μορφής για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα και η πολιτική αυτή χρειάζεται να προωθηθεί καλύτερα ώστε οι επιχειρήσεις ενεργά να τις εφαρμόσουν και θα πρέπει να δούμε και πόσο εταίρος και πόσο πελάτης τα βλέπουν αυτά σε αυτές τις επιχειρήσεις γιατί η στήριξή τους είναι πολύ σημαντική για την εφαρμογή του συστήματος. Θα ήθελα επίσης για μια ακόμα φορά να τονίσω την ε, άριστη εργασία των συντακτών της εισήγησης θεωρώ ότι θα πετύχουμε μια κοινή έκφραση και συνένεση πάνω σε αυτό. Ναι, και εγώ έχω μια άποψη. Πολλές επιχειρήσεις ευρωπαϊκές ε, συμμετέχουν ιδιαίτερα στην στήριξη υποψηφίων στις ΗΠΑ ε, είτε για τον πρόεδρο και για άλλους υποψηφίους στη Βουλή ή στη Γερουσία και τώρα για την στήριξη αυτών των υποψηφίων στις πολιτείες υπάρχει μια διαφάνεια και υπησέρχεται στα σχετικά αυτά πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, γιατί βλέπουμε διάφορες ισχυρές επιχειρήσεις να είναι υπέρ υποψηφίων που είναι υπέρ του κλίματος ας πούμε να δούμε τι γίνεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πώς θα μπορέσει η κοινή γνώμη να τα παρακολουθήσει. Ο κύριος Παλάθιο από πλευράς Επιτροπής μήπως θα ήθελε να μας πει κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Μερικά σχόλια θα ήθελα να κάνω σε σχέση με τη γνωμοδότηση αλλά και σε σχέση με τη συζήτηση που άκουσα σε σχέση με την ανακοίνωσή μας του 2011, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε μία νέα θέση ε, σε σχέση με το κατά πόσο το ΣΕ είναι ε, υποχρεωτικό ή εθελοντικό, θεωρώντας ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στην κοινωνία. Δεν έχει σημασία κατά πόσο είναι υποχρεωτικό ή εθελοντικό. Ε, μιλάμε για τις πιθανές συνέπειες και τη δυνατότητα ε, που έχουν οι επιχειρήσεις να επηρεάσουν την κοινωνία. Θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε μέσω της εταιρικής κοινωνικής ε, ευθύνης τις θετικές συνέπειες και να ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές. Αλλά επιστρέφοντας στα σημεία που αναφέρει και η γνωμοδότηση δεν λαμβάνει υπόψη κάποιες από τις πρόσφατες εξελίξεις ε, στην ε, χάραξη πολιτικής από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι κάτι το οποίο όντως αναφέρεται στις τελευταίες συμφωνίες με την Κολομβία του Περού, το Καριφόρουμ, ούτως ή άλλως λοιπόν έχουμε συμπεριλάβει την πτυχή αυτή. Επίσης, στις τελευταίες μας ανακοινώσεις μας για τις επενδύσεις το 2011 αλλά και για την ανάπτυξη του εμπορίου αναφερόμαστε σε αυτό το θέμα διαπραγματευόμαστε ρήτρε ε, που συμπεριλαμβάνουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη στις, ε, ελεύθερες εμπορικές, ε, στις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και θα το κάνουμε και στις επενδυτικές συμφωνίες που θα προκύψουν. Όσον αφορά τώρα τη ρήτρα αυτή, Θα ήθελα να πω ότι προτείνουμε τους, τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΣΑ ε, για ε, το θέμα αυτό ε, σε σχέση με την εφαρμογή κυρίως, με τα μέτρα εφαρμογής. Υπάρχουν μάλιστα και σημεία επαφή στις διάφορες χώρες μέλη. Ε, δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι θέλουμε να συμπεριλάβουμε τόσο λεπτομερές, ε, τόσο τέτοιο επίπεδο λεπτομεριών στις ε, συμφωνίες μας. Μπορούμε να παραπέμπουμε στις κατευθυντήριες γραμμές του ΩΣΑ, που κατά τη γνώμη μας είναι η πιο, το πιο περιεκτικό μέσο που υπάρχει για το θέμα της εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρθηκε το Global, το Global Compact, η Διεθνή Οργάνωση Εργασία. Όμως ε, για μας οι κατευθυντήριες γραμμές ε, του ΩΣΑ είναι πολύ σημαντικές γιατί συμπεριλαμβάνουν έναν μηχανισμό εφαρμογής ε, χωρίς να χρειάζεται υποχρεωτικά να προσθέσουμε επιπλέον διατύπωση στις συμφωνίες μας. Όσον αφορά τώρα το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ, είναι ένα μέσο συμφωνίας μεταξύ κυβερνήσεων. Δεν αφορά ε, λήψη αποφάσεων από εταιρείε. Δεν το συμπεριλαμβάνουμε λοιπόν αυτήν την, την εταιρική κοινωνική ευθύνη ε, στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ω τέτοιο, αλλά υπάρχουν ούτω ή άλλω τέτοιε πτυχέ. Όλα αυτά που κάνουμε πρέπει να είναι και συμβατά με τον ΠΟΕ και θα συμπεριλάβουμε βέβαια τις πτυχές αυτές, όμως από την άλλη πρέπει να υπάρχει και ένας μηχανισμός που να είναι ε, συμβατός με τον ΠΟΕ. Όσον αφορά τώρα την ε, νομική συνεργασία και την αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη, Πιστεύουμε ότι αυτό κάπως υπερβαίνει τις ε, προσδοκίες μιας εμπορικής συμφωνίας και των αποτελεσμάτων αυτή. Αυτής είναι τμήμα της εξωτερικής πολιτικής ή της αναπτυξιακής πολιτικής ενδεχομένως, όχι όμως της εμπορικής πολιτικής. Συμφωνούμε με το στόχο βέβαια του να υπάρξουν τέτοιοι μηχανισμοί, αλλά δεν θεωρούμε ότι οι εμπορικές συμφωνίες είναι το σωστό μέσο για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά. Όσον αφορά τώρα το θέμα της ισορροπίας μεταξύ την, ε, της προστασίας των επενδυτών και της κρατικής ενίσχυσης, ε, είναι σημαντικό τμήμα της επενδυτικής πολιτικής. Έχουμε σκοπό να το συμπεριλάβουμε και εμείς ε, στις επόμενες επενδυτικές μας συμφωνίες. Θα υπάρχουν ρήτρες όσον αφορά το δικαίωμα ρύθμισης, ε, να εξασφαλίσουμε δηλαδή ότι διατηρείται το δικαίωμα αυτό ε, στη, στο πλαίσιο των ε, διμερών επενδυτικών συμφωνιών ε, και θα προσπαθήσουμε επίσης να προωθήσουμε τη δέσμευση των επιχειρήσεων για τα υψηλότερα πρότυπα επαγγελματικής, ε, ε, επιχειρηματικής διοντολογίας. Και ένα τελευταίο θέμα που θα ήθελα να θέσω σε σχέση με την τροποποίηση της λογιστικής οδηγίας και της οδηγίας περί διαφάνειας. Δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ συνάδελφος Γενικής Διεύθυνσης Μάρκετ. Ε, όμως αυτό που ξέρω είναι ότι η συγκεκριμένη Γενική Διεύθυνση αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται έναν κανονισμό δεν ξέρω ποιο, θα είναι το τελικό καθεστώς αυτού του κειμένου, αλλά αφορά ε, ε, τα, οικονομικά και ειδικότερα του ενοποιημένου λογαριασμού και τη σχετική οδηγία. Οι πρωτοποποιήσει αυτέ θα συμπεριλάβουν βεβαίω στοιχεία ε, μη οικονομική λογοδοσία και οικονομική λογοδοσία. Είναι κάτι το οποίο έχει δρομολογηθεί αυτέ τι μέρε υποθέτω ότι θα γνωστοποιηθεί σύντομα ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι τροποποιήσεις αυτές δηλαδή θα γνωστοποιηθούν σύντομα. Και είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να έπρεπε να ληφθεί και αυτό υπόψη στη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής, ο κύριος Λάγκε. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τους αδέλφους για τα σχόλια και τη συμβολή του στην έκθεση. Θα τη βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο πιστεύω. Μπορούμε να διαπιστώσουμε νομίζω ότι ακολουθούμε την ίδια κατεύθυνση και ενισχύουμε τον τομέα των ευρωπαϊκών αξιών για τις δραστηριότητες και τις διεθνείς των ευρωπαϊκών επιχειρήσουν. Έτσι ώστε να μην λησμονούν ε, τι ε, ανθρώπινε αξίε όταν δραστηριοποιούνται εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να διατυπώσω κάποιε παρατηρήσει αλλά και ερωτήσει. Εσείς λέτε ότι δεν χρειάζεται καν έκθεση, τα έχετε καλύψει όλα. Εγώ όμως έχω ριζικά αντίθετη γνώμη και πιστεύω ότι η κατάσταση της εταιρικής ε, κοινωνικής ευθύνης, τουλάχιστον στις ε, εμπορικές σας συμφωνίες, όταν καταγράφεται αναφέρεται μόνο ως μία βούληση για προώθηση της ΕΚΕ. Τίποτε πιο συγκεκριμένο. Άρα χρειάζεται περισσότερη βελτίωση στη δική σας, ε, στις δικές σας συμφωνίες. Η την ενσωμάτωση στο γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων και γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων συν θα πρέπει να δούμε πώς με σε αυτούς όρους μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό και βέβαια πώς θα αντιδράσουν και θα συμπεριφερθούν οι εταιρείε. Τελευταία παρατήρηση και το ζήτημα της διαφάνειας στις ε, μηνιαίες ε, και ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων των επιχειρήσεων. Πολύ ωραίο είναι αυτό, μακάρι να πραγματοποιηθεί. Θα περιμένουμε βεβαίως να δούμε τις προτάσεις αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να τις αξιολογήσουμε. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω και το εξή. Στην ανακοίνωση. Βλέπω μια σειρά 13 συγκεκριμένων ε, διαβημάτων, εάν δεν απατώμε, και ενώ έχει περάσει ένας χρόνος, γιατί νομίζω πέρσι τον Οκτώβριο δημοσιεύτηκε αυτή η ανακοίνωση, Εκεί που λέτε επί παραδείγματι ότι τα επενδυτικά κεφάλαια και τα χρηματοοικονομικά Ινστιτούτα χρηματοπιστωτικά Ινστιτούτα θα πρέπει να καταγράφουν ε, τις δραστηριότητες προς, ως προς την ε, δεοντολογία και την ε, τήρηση των κανόνων αυτής στις εκθέσεις πεπραγμένων. Το κάνατε όντως αυτό, συνέβη αυτό που λέει η ανακοίνωση. Επίσης, Λέτε κάπου αλλού ότι για τις μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να υπάρξει στο 2014 υποχρέωση για την τήρηση των προδιαγραφών ε, ΕΚΕ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο μέχρι το 2014, άρα είτε πρόκειται για το 26.000 ίζο, είτε πρόκειται για το Global Compact, είτε για οποιασδήποτε άλλες διατάξεις και προδιαγραφές του ΩΣΑ. Θα ήθελα να μου πείτε αν βλέπετε κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις της Ευρώπης οι οποίες προχωρούν προς την κατεύθυνση αυτή για να τηρήσουν τις εν λόγω προδιαγραφές, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Και επίσης ένα άλλο από τα 13 μέτρα που είχατε προτείνει ήταν τα κράτη-μέλη έως το 2012, το οποίο λίγοι όσο πω θα είχαν εισαγάγει κατευθυντήριες γραμμές προαγωγής ε, της εταιρική κοινωνικής ευθύνης και θα ζητούσατε, θα, θα προβλέπατε μάλλον μια διαδικασία peer review, δηλαδή επαλήθευση από τους εταίρους ε, συμπεριφορά συμπεριφοράς των κρατών μελών ως προς την εισαγωγή αυτών διατάξεων. Μέχρι, μέσα στο 2012 έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, ακούσαμε κάποιες ερωτήσεις, μήπως θα θέλατε να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ σε σχέση με τα επενδυτικά ταμεία και το τι γίνεται σε σχέση με την ε, ε, εταιρική κοινωνική ευθύνη. Έχουμε ευθυγραμμιστεί με τη δουλειά του ΩΣΑ, δηλαδή την ανάπτυξη των κατευθυντηρίων γραμμών για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, δεοντολογία δηλαδή για ε, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Έχει ξεκινήσει αυτή η δουλειά η ιδέα είναι να καλύψουμε όλες τις πτυχές ΕΚΕ στις διάφορες συναλλαγές των διαφόρων χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων και τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων αλλά και τους διαχειριστές άλλων επιχειρηματικών μοντέλων. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν να χαρτογραφήσουν στον ΟΣΑ τα διάφορα επιχειρηματικά ε, μοντέλα τα οποία χρειάζονται περισσότερο, περισσότερες ε, κατευθυντήριες ε, γραμμές και οι πτυχές ε, του χρηματοοικονομικού κλάδου ήδη λαμβάνονται υπόψη, ε, λαμβάνεται υπόψη και η εταιρική κοινωνική ευθύνη Υπάρχουν και οι προδιαγραφές του ΟΗΕ για τις υπεύθυνες επενδύσεις, ε, τις έχουμε προσυπογράψει και αυτές. Ε, έχουμε και εμείς κάποιες αρχές ε, για, την, για τα σωστά οικονομικά, όμως προσπαθούμε να τα καταγράψουμε όλα αυτά και να τα θέσουμε, να τα θέσουμε στο πλαίσιο της, των επιχειρήσεων για να δούμε τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή θα συνεχίσει ε, την παρακολούθηση των εργασιών του ΩΣΑ στον τομέα αυτό. Όσον αφορά τώρα τις θεσμεύσεις ε, του, για το σχέδιο δράσης ε, της ανακοίνωσης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, Έχουμε τετραμηνιές ή εξαμηνιές εκθέσεις ε, για τα θέματα αυτά. Βέβαια, οι συνάδελφοι της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων ασχολούνται κυρίω με αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά θα υποβάλουν και σε εμά μια έκθεση όλων αυτών των στοιχείων, ε, Ούτω ή άλλω ε, και, ούτως ή άλλως είναι αντικείμενο και μιας αξιολόγησης ομοτήμων. Ελπίζουμε σύντομα να ξεκινήσουμε τις σχετικές δραστηριότητες. Με τα κράτη-μέλη συνεργαζόμαστε, παρα, Έχουμε τις ομάδες κρατών μελών που παρατηρούν τις διάφορες πτυχές της εταιρική κοινωνικής ευθύνης. Έχουμε την ομάδα υψηλού επίπεδου η οποία συνέρχεται κάθε έξι μήνες και θα έχουμε και μία συνάντηση της ομάδας αυτής τους ερχόμενους μήνες. Θα γίνει επίσης και η συνάντηση του φόρουμ ε, των εμπλεκομένων φορέων Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο πλαίσιο της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής. Όσον αφορά τώρα τις υπόλοιπες δραστηριότητες ε, που προβλέπει η ανακοίνωση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, από ό,τι κατάλαβα πηγαίνουν καλά ε, τα πράγματα. Το θέμα της οικονομικής λογοδοσίας, ναι, έχετε δίκιο, αυτό καθυστερεί λιγάκι, αλλά από ό,τι κατάλαβα ούτως ή άλλως έχουμε κανόνες στη διάθεσή μας ε, και ελπίζουμε σύντομα να τους μοιραστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Είστε ικανοποιημένο. Μάλιστα, προθεσμία υποβολής τροπολογιών 14 Νοεμβρίου στις 6 ε, το απόγευμα. Ε, autre Επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξής μας είναι το 10 για την, ε, τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες, εμπόριο και ανάπτυξη βασισμένη σε επενδύσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Το και είναι η συγγετριά μας, από ό,τι κατάλαβα εκπροσωπείται από τον Μάριο Νταβίδ σήμερα. Γνωρίζετε ότι συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή Ανάπτυξης σε αυτό το θέμα. Πριν δώσω το, το λόγο στον ε, εισηγητή, να γνωρίζετε ότι θα υπάρξει και μία παρουσίαση από τον κύριο Καρίμ Νταού, ο οποίος προέρχεται από τον ΟΣΑ και ο οποίος ε, ασχολείται με το θέμα των επενδύσεων στην Αφρική του ε, στον ΟΣΑ μπορεί και εκείνο ε, να δώσει ε, στοιχεία για τη συζήτησή μας. Ο ε, Αλμπέρτο μου είπε ότι Το γεγονός ότι είναι εδώ ο εκπρόσωπος του ΟΣΑ δικαιολογεί της, ε, τη συνοχή μεταξύ των εργασιών των δύο επιτροπών, της Διεθνούς Εμπορίου και της Ανάπτυξης. Ε, θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στον ε, Μάριο για να μας πει περισσότερα. Ναι. Δεν λέτε τίποτα για τη συνοχή του ΕΛΚ πάνω σε οποιοδήποτε θέμα. Τέλος πάντων, το ίδιο και για όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Δεν διαφέρουμε από τις υπόλοιπους, έτσι. Να ακούσαμε το σχόλιο του Πρόεδρου. Ο μιλητής λέει ευτυχώς. Το και σοφή στα συγγνώμη λυπάται που είναι απούσα σήμερα. Εγώ θα εκφράσω όλα αυτά και επίσης να σας πω την διαθεσή σας για να συζητήσετε την, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής για το θέμα αυτό. Κάτι για τη διαδικασία. Όπως την αναφέρατε εσείς κύριε Πρόεδρε, η Τόκια τι να πει ότι συντάσσει ένα κείμενο σχετικά με αυτή την ανακοίνωση του Ιανουαρίου του 2012 που είναι η βάση για την έκθεσή σας, είναι κοινό το χρονοδιάγραμμα και ε, βάσει του άρθρου 50 εργάζονται οι δύο επιτροπέ και υπάρχει μια κατανομή αυστηρή ακριβώ των αρμοδιοτήτων και θέλουμε η συγγήτρια, θέλει η συγγήτρια να σεβαστούμε όλοι μα στην ίντα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για το εργαλείο συνεργασία την ανάπτυξη γιατί είναι αποκλειστική αρμοδιότητα ε, τη επιτροπή ανάπτυξη. Ε, έχουμε όμω μια αρμοδιότητα αποκλειστική για τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών και οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με το εμπόριο. Και εδώ με τι υποχρεώσει αυτέ. για τη σύνταξη, έτσι διάφορα θέματα. Η συγγήτρια δεν μπόρεσε να εξετάσει όλα όσα δίνουν μια απάντηση σε αυτά τα κύρια σημεία που καθοδηγούν την εργασία της, δηλαδή πώς το εμπόριο και η επένδυση θα μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά την ανάπτυξη των χωρών των ε, αναδειωμένων. Και εδώ δεν είναι αυτό σκοπό το εμπόριο, αλλά επίση συμφωνούμε ότι εάν συνοδεύεται από συμπληρωματικά μέτρα, εάν σέβεται το ρυθμό ανάπτυξη των, των εμπορικών μα εταίρων και τι τις αρχέ εξωτερικέ τη Ένωση, τότε θα μπορούσε να έχει μια θετική επίδραση. Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες οι αναπτυσσόμενες καθορίζουν τη βάση της ανάπτυξης, στην πολιτική τους και υιοθετούν μέτρα που προτείνουν οι ανεπτυγμένες χώρες και δημιουργεί απασχόληση σε αυτές τις χώρες σύμφωνα με τη συγκήτρια αποτελεί σημαντικό σημείο το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Το 2 θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το πώς επηρεάζει η οικονομική κρίση την προσφορά βοήθειας ε, στις ε, ανεπτυσσόμενες χώρες και όλα αυτά έχουν τρεις επιπτώσεις. Πρώτα απ' όλα για το συνολικό ύψος ε, αφού το συνολικό ύψος αυτής της χρηματοδοτικής βοήθειας μειώνεται, οι εταίροι θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματικότητα τα υπάρχοντα κονδύλια μέσω καλύτερου συντονισμού ανάμεσα στου ε, διάφορου παράγοντε. και αυτό, πάνω σε αυτό θα μπορούσε να προσφέρει προ τη προστιθέμενη αξία Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά θα πρέπει να εγκαταλείψει την ιδέα μια σκέτα οικονομική βοήθεια και να προχωρήσει σε μια τεχνική ας πούμε βοήθεια στο εμπόριο που έχει διάφορα πλεονεκτήματα, δεν επηρεάζει τον προπολογισμό των αναπτυγμένων χωρών και επηρεάζει τα πράγματα χρονικά μακρύτερα και επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι αρμοδιότητες και το προσωπικό για να βοηθούν οι λιγότερο επτυγμένες χώρες ε, με την ένταξή τους στον ΩΣΑ και να βοηθούν οι χώρες αυτές οι οποίες ζητούν την ένταξη να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία τους ε, και στο ε, ε, οργάνωση εμπορίου με καινούριο κατάλληλο τρόπο. Επίσης, ένας καινούριος τρόπος χρηματοδότησης καταλαβαίνει η κυρία Τόκια ότι τα μικροπιστώσεις είναι μέθοδοι που έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους. Αλλά να δούμε για τα μεγάλα διαφορετικά έργα είναι αποτελεσματικά. Η συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου φορέα και η τριμερή συνεργασία με τις χώρες ε, και του Βορρά και του Νότου είναι συγκεκριμένες Και τώρα για τις διαπραγματεύσεις των εμπορικών συμφωνιών διμερών ή περιφερειακών θα πρέπει να διαφέρουμε από την παραδοσιακή λογική, θα πρέπει να είμαστε υπέρ της ανάπτυξης και το πώς θα συμπεριληφθούν στο εμπορικό παγκόσμιο σύστημα αυτές οι χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει υπόψη μας το πώς θα επηρεάσει αυτή η συμφωνία τη ζωή στο μέλλον και με βαθιά επίδροση για να δούμε για τα τέλει ακριβώς αν θα εξαφανιστούν ή όχι και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προτείνει μέτρα κάτι περισσότερα από μια ε, ρύθμιση διευθέτηση στον τομέα του εμπορίου. Εάν η συγγήτρια βέβαια παρόλο που συμφωνεί με τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ανακοίνωσή της ε, λυπάται όμως ε, γιατί δεν προχωράει περισσότερο η Επιτροπή πέρα από μια ενημέρωση στρατηγικής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2002. Εκφράζει τη λύπη της γιατί η Επιτροπή δεν βλέπει το νέο ρόλο που παίζουν ε, οι αναδυόμενες χώρες στο διεθνές κοινικό ξεκινώντας από τη βοήθεια στο εμπόριο και επίσης θα πρέπει να υπάρξει βοήθεια που να έχει σχέση με τις αναδυόμενες και όχι τις ανεπτυγμένες χώρες. Ε, δυστυχώς υπάρχουν προοπτικές που θα πρέπει να αποφευχθούν και η συγκήτρια εκφράζει τη λύπη γιατί η Επιτροπή δεν δείχνει την αλεπίδραση των οικονομιών μας αμοιβαία. Θα μπορούσαμε να δούμε ακριβώς ε, στον τύπο ότι η Καντών ε, πλήττεται από την κρίση της ζώνης ευρώ γιατί είναι στραμμένη η εξαγωγή της προς εμάς και για να δώσουμε τις κατάλληλες αποτελεσματικές λύσεις θα πρέπει να αποδείξουμε ότι μας δεκατέχει περισσότερος ρεαλισμός και υπέρ των χωρών που απολαμβάνουν τις βοήθειάς μας. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για την προσοχή και οπωσδήποτε τις παρατηρήσεις σας ακριβώς θα τις μεταβιβάσω στην συνάδελφο την κυρία Τοκία Σάιφη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν δώσω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές ε, να ακούσουμε την ε, παρουσίαση του ΩΣΑ. ώστε να έχουμε υποφεληθεί πλήρως ε, και από την εξαιρετική παρουσίαση του εκπροσώπου της εισηγήτριάς μας, αλλά και του κυρίου Νταού. Ε, σας δίνω το λόγο για 10 λεπτά και μετά θα ακούσουμε αντιδράσεις και σχόλια ε, των μελών της Επιτροπής μας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Θα κάνω την παρουσίασή μου στα αγγλικά. Ευχαριστώ. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα όλους να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του ΟΟΣΑ γιατί μας προσκαλέσατε να ε, συμβάλλουμε κι εμείς σε αυτή την ενδιαφέρουσα ε, συζήτηση για την επένδυση για την ανάπτυξη. Εγώ είμαι διευθυντής της Επιτροπής της Επενδυτικής του ΟΟΣΑ που επικεντρώνεται κυρίως στις, ε, στην σχέση της επένδυσης με την ανάπτυξη. Πριν όμως ε, πω ορισμένα πράγματα για τι εργασίε του ΩΣΑ στον τομέα αυτό, θα ήθελα για ένα λεπτό να σας ε, αναφερθώ στην ε, άποψή μα εντυπωσει μας για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα σχόλια του εισηγητή. Καταρχά χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέματα όπως το εμπόριο το συνδέει σε μεγάλο βαθμό με την ανάπτυξη γιατί θεωρούμε ότι είναι συμπληρωματικά ε, γιατί η επένδυση ε, για την αναβάθμιση της παραγωγής ε, των χωρών αλλά και ορισμένων αλυσίδων προϊόντων μπορεί να είναι πραγματικά πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη των αναπτυσσομένων χωρών. Η σχέση λοιπόν επενδύσεων και ανάπτυξης είναι πάρα πολύ σημαντική στην αναπτυξιακή διαδικασία. Όσον αφορά τώρα την ανακοίνωση και την έκθεση εμείς δεν έχουμε καμία ιδιαίτερη αντίρρηση. Θεωρούμε ότι και τα δύο πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα θέλαμε απλώς να προσθέσουμε κάποια σχόλια τα οποία θα μπορούσαν να συμπληρώσουν ε, τα ε, δύο αυτά κείμενα. Πρώτον πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε το ρόλο της ε, αναπτυξιακής βοήθειας, από κοινού με τις επενδύσεις, όμως είναι καινοτόμος ο ρόλος που μπορεί να παίξει ε, η αναπτυξιακή βοήθεια για την ανάπτυξη πολιτικών σε αναπτυσσόμενες χώρες, ε, για την ενίσχυση και τη βοήθεια των αναπτυσσομένων χωρών, ε, ας πούμε, σε περιβαλλοντικές πτυχές ας πούμε τον τομέα των υποδομών ε, που είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη μιας ικανότητας προσφοράς ε, είτε μπορεί καλή, κανείς να την υποστηρίξει με υλική υποδομή ή μπορεί με διάφορες πολιτικές μέσω επενδύσεων να την, ε, να την προωθήσει. Νομίζουμε ότι το δεύτερο είναι εξίσου σημαντικό με το πρώτο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ο ρόλος της βοήθειας, ο καινοτόμος ρόλος σε σχέση με την ενίσχυση της ε, πολιτικών, ανάπτυξης πολιτικών των αντισωμένων χωρών είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι κάτι το οποίο ε, αναφέρεται και στην έκθεση και στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύουμε επίσης ότι το γεγονός ότι οι επενδύσεις ε, ε, εξετάζονται περισσότερο ως συνεισφορά σε αυτό το τομέα είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ με τις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά την ενίσχυση του, τομέα της προσφοράς. Ε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την οικοδόμηση των ικανοτήτων ε, ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων σε αναπτυσσόμενες χώρες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα ως προς αυτό. Ε, συμφωνούμε και με την έκθεση και με την ε, ανακοίνωση της Επιτροπής, οπότε καλό είναι να περάσω τώρα στην εργασία του ε, ΩΣΑ ε, στον τομέα της ανάπτυξης και της επένδυσης. Έχουμε τώρα ένα νέο φορέα, ένα νέο φορέα που λέγεται Συμβουλευτική Ομάδα Επένδυσης και Ανάπτυξης, που συγκεντρώνει εκπροσώπους της Επενδυτικής Επιτροπής του ΩΣΑ, αλλά και της Αναπτυξιακής Βοήθειας, Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας, και αυτές οι δύο είναι υπεύθυνε για για την, επεν, για την ε, εποπτεία της εργασίας μας όσον αφορά τις επενδύσεις, τον τομέα των επενδύσεων. Θέλουμε λοιπόν έτσι να κινητοποιήσουμε τη συλλογική γνώση ε, ορισμένων κοινοτήτων ε, ε, ε, υπεύθυνων πολιτικών σε αυτούς τους δύο τομείς. Είναι πολύ σημαντικό γιατί οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας μπορεί να ενθαρρύνουν τους συναδέλφους τους από την Αναπτυξιακή Συνεργασία συνεργασία και από άλλους φορείς ε, να ευθυγραμμίσουν, ε, να συμπεριλάβουν δηλαδή το τομέα των ε, επενδύσεων στις σχέσεις τους με τις ενδιαφερόμενες χώρες τέσσερις διόδους εργασιών. Έχουμε την ε, ανοιχτή και ε, ε, διαφανή πολιτική για την επένδυση, την ενίσχυση της υπεύθυνη επιχειρηματικής συμπεριφοράς, την ενίσχυση της αμοιβαία ωφέλειας για τις διεθνείς επενδυτικές συμφωνίες και τις καλύτερες στατιστικές διεθνών επενδύσεων. Όλα αυτά είναι αλληλοσυμπληρούμενα ε, για το πρώτο, ε, την ανοιχτή και διαφανή ε, πολιτική, ένα πλαίσιο διαφανούς και ανοιχτής πολιτικής για την επένδυση. Ε, υπάρχει η πτυχή της χώρας προέλευσης ας πούμε αλλά και της χώρας υποδοχής της επένδυσης. Ε, προσπαθούμε ειδικότερα στο επίπεδο της χώρας ε, υποδοχής να βοηθήσουμε τις σχετικές υποδομές. Προσπαθούμε με διάφορους τρόπους που θα σας πω πολύ σύντομα να το πετύχουμε αυτό και σε κρατικό επίπεδο προσπαθούμε να υπάρξει διάλογος μεταξύ όχι μόνο των χωρών του ΩΣΑ αλλά και των αναδειωμένων ανεπτυγμένων οικονομιών ε, για να υπάρξει ένα ανοιχτό επενδυτικό πλαίσιο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις αναπτυσσόμενες χώρες σε ένα πλαίσιο στο οποίο αποτελούν όλο και περισσότερο ε, αντικείμενο επενδύσεων και συνεπώς μπορεί να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό από τον ε, επενδυτικό προστατευτισμό των χωρών του ΩΣΑ. Όσον αφορά τώρα την προώθηση των, της υπεύθυνη επιχειρηματικής συμπεριφοράς, ε, το αναφέρατε και στη συζήτηση εδώ σήμερα. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές για το θέμα αυτό και ενημερώθηκαν το 2011 από τον ΩΣΑ δύο βασικές καινοτομίε εισήχθησαν. Πρώτον, το κεφάλαιο για τα, ανθρώπινα δικαιώματα έχει ενισχυθεί πολύ και δεύτερον, και είναι νομίζω σημαντική εξέλιξη, μία ε, ένας κώδικας συμπεριφοράς ε, που έχει συμπεριληφθεί ε, στην εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών. Όχι μόνο δηλαδή εστιάζουμε στην ευθύνη του κράτους προ, υποδοχής, ε, προκυ... Ε, συγγνώμη, προέλευσης ως προς τη συμπεριφορά των πολυεθνικών εταιριών που πηγαίνουν σε μια χώρα. Υπάρχει και ενισχυμένος διάλογος με τις επιχειρήσεις, με τον επιχειρηματικό κλάδο, ώστε να ε, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ε, αρνητικών συνεπειών ε, ε, σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό επίπεδο ή και βάσει άλλων προτύπων με τα οποία πρέπει να συνάδουν πλέον η, τα οποία πρέπει να συνάδει η επιχειρηματική συμπεριφορά. Υπάρχει λοιπόν συνεχής διάλογος για τα θέματα αυτά, ώστε να μπορούμε να συγκεράσουμε των δύο χωρών τα συμφέροντα της χώρας προέλευση επένδυσης αλλά και της χώρας υποδοχής και επίσης καλύτερες, καλύτερες στατιστικές ε, σε διεθνές επίπεδο. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις χώρες αυτές ε, στην ικανότητά τους να έχουν στατιστικές που μπορούν να ε, ενημερώνουν τις πολιτικές τους. να σας πω ποιο είναι το βασικό μας μέσο για την επενδυτική πολιτική, ε, που είναι το πλαίσιο πολιτικής για την επένδυση, το PFI. 30 χώρες του ΩΣΑ και 30 ε, χώρες που δεν είναι μέλη του ΩΣΑ για μια περίοδο 5 ετών ε, έχει χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον 30 χώρες, περίπου 30 χώρες κατά κύριο λόγο αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιούμε για να τις βοηθήσουμε να αξιολογούν και να μεταρρυθμίζουν το πλαίσιο επένδυσης τους, το επενδυτικό τους πλαίσιο. Δεν αφορά μόνο την επενδυτική πολιτική, αλλά αφορά όλους τους τομείς πολιτικής που έχουν συνέπεια στον επιχειρηματικό κλάδο, ανταγωνισμό, υποδομές, χρηματοοικονομικές αγορές, ε, ε, εταιρική διακυβέρνηση κλπ ε, είναι ζητήματα τα οποία υπεύθυνοι χάραξη πολιτική πρέπει να τα λάβουν υπόψη. Δεν είναι όμω υποχρεωτικά. Προσπαθούμε να προωθήσουμε την συνοχή των πολιτικών ε, των επενδυτικών και προσπαθούμε επίσης ε, ε, κάποιους δημόσιους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για το εμπόριο για παράδειγμα να τους βοηθήσουμε να συμπεριλάβουν ένα πλαίσιο επενδυτικό το οποίο να είναι όσο πιο συνεκτικό και περιεκτικό γίνεται. Εκτός λοιπόν από την ε, ενίσχυση των αναπτύξεων αναπτυξωμένων χωρών στην προσπάθειά τους ε, να αναβαθμίσουν το διεθνή τους ρόλο. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν ε, κάποια μεγαλύτερη εξειδίκευση σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Υπάρχουν χώρες ε, για τις οποίες η ανάπτυξη των υποδομών είναι προτεραιότητα, ενώ για άλλες χώρες, για παράδειγμα ο γεωργικός τομέας είναι ένας βασικός κινητήριος μοχλός ανάπτυξης. Άρα λοιπόν έχουμε διάφορα τομεακά εργαλεία που προκύπτουν από το PFI και που δίνουν τη δυνατότητα δυνατότητα στις χώρες αυτές ε, να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν το δυναμικό τους, το επενδυτικό το τομείς αυτούς. Έχουμε λοιπόν ε, ε, τις αρχές για την σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, στον τομέα των υποδομών για παράδειγμα. Οι πράσινες επενδύσεις είναι επίσης βασική για μας, βασικό μέλημα για μας, Έχουμε συμπεριλάβει ειδικά κεφάλαια στο PFI για τις πράσινες επενδύσεις, ε, πώς είναι δυνατόν δηλαδή το δυναμικό το επενδυτικό να εξελιχθεί σε μια πιο πράσινη ε, κατεύθυνση και έχουμε επίσης και σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών ε, για την καθαρή ενέργεια ε, και μιλάω για περίπου το ίμιση της Αφρικής. Ε, πρόκειται για ένα εργαλείο που εξετάζει πώς θα επιστρατευτούν επενδύσεις προς την κατεύθυνση της καθαρής ενέργειας και έχουμε επίσης και ένα πλαίσιο πολιτικής για τη γεωργία Μπουργκίνα Φάσο, Ινδονησία, Τανζανία και θα συνεργαστούμε σύντομα και με την ε, Μιανμάρ για τον τομέα αυτό, ώστε αυτές οι χώρες να μπορούν ε, να ε, προωθήσουν επενδυτικές ροές στον γεωργικό τομέα. Και βεβαίως η υπεύθυνη επιχειρηματική πολιτική, ανέφερα ήδη τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Ίσως αυτό που θα έπρεπε να προσθέσω είναι το εξής, ότι εκτός από την αντιμετώπιση του ζητήματος της ε, υπεύθυνη συμπεριφοράς των επιχειρήσεων ε, ε, σε επίπεδο προέλευση επενδύσεων, θέλουμε να δούμε και πώ οι χώρε υποδοχή μπορούν να ενισχύσουν το σύστημα διακυβέρνηση του, διαχείριση των εταιριών, να δούμε δηλαδή το νομικό και το ρυθμιστικό πλαίσιο για την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά. Δεν αφορά δηλαδή μόνο τις προσδοκίες τις κοινωνικές, αλλά έχει να κάνει και με το νομικό και ρυθμιστικό ε, πλαίσιο τις ε, δεσμευτικές απαιτήσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, τα κοινωνικά πρότυπα, τα πρότυπα καταπολέμησης της διαφθοράς κλπ. Εκτός από την ανάπτυξη εργαλείων και τη συνεργασία με τις χώρες για την επενδυτική πολιτική, επίσης προωθούμε έναν παγκόσμιο διάλογο για το θέμα αυτό, και έχουμε και κάποια ε, στοιχεία τα οποία προσπαθούν, ε, προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα της συνεργασίας ε, της επενδυ, στην επενδυτική πολιτική. Έχουμε ένα φόρουμ κάθε δύο χρόνια για το θέμα αυτό και όπως είπα και προηγουμένως ε, μας δίνει τη δυνατότητα το φόρουμ αυτό να καταπολεμήσουμε τον επενδυτικό προστατευτισμό σε, μια, σε ένα ευρύτερο οικονομικό ε, ε, πλαίσιο, αλλά επίσης προσπαθούμε να ε, ενθαρρύνουμε τη συνομιλία των αναδειωμένων χωρών με τους ενδεχόμενους επενδυτές. Έχουμε... Επίσης έχουμε συνομιλίες και συνεννόησεις με τις αφρικανικές χώρες, με την νοτιοαφρικανική κοινότητα, με την ΑΣΕΑΝ της ΣΑΤΚ ε, Αναπτυξιακή Κοινότητα της Νότια Αφρικής και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη γιατί έχουμε συνοηθεί με τη ΣΑΤΚ για έναν πλαίσιο συνεργασία για τι επενδύσει τη ΣΑΤΚ που χρησιμοποιεί ω σημείο αναφορά το PFI, το πλαίσιο αναφοράς, το πλαίσιο πολιτικής για τις επενδύσεις. Και επίσης έχουμε χώρες ε, γειτονικέ πολλές φορές, οι οποίες μεταξύ τους ε, βρίσκονται σε ανταγωνισμό για το ποια θα δώσετε τις πιο, τα πιο χαμηλά ε, ποσοστά. Μια περιφερειακή λοιπόν συνεργασία, πολύ σημαντική, πολύ ενδιαφέρουσα και με αυτά τα ολίγα τέλειωσα την παρουσίασή μου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Merci. Σας ευχαριστώ κύριε Ντάου για όσα μας είπατε, ιδιαίτερα χρήσιμα και γιατί μας εξηγήσατε την εργασία του ΩΣΑ πάνω στο θέμα αυτό. Η σκιώδηση συγγήτρια Μαρία Βαντία. Καλημέρα Πρόεδρε, να ευχαριστήσω για την εξήγηση του ΩΣΑ, για όσα λέμε τώρα και πραγματικά μας βοηθά ιδιαίτερα για να προσανατολιστούμε ακριβώς ε, και πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε τις εργασίες μας. Η άποψή μου για την αρκίνωση της Επιτροπής είναι ότι απαιτείται πραγματικά και να ασχοληθούμε για να δούμε και την τελευταία με την ε, ανάπτυξη του από το 2002 και μετά, γιατί οι αναπτυσσόμενες χώρες, αυτά που είπαμε, θα πρέπει να αναθεωρηθούν και σαν ομοιόμορφη ομάδα μεταβλήθηκε λόγω των οικομικών αλλαγών και την αλλαγή του διεθνού κοινικού και ορισμένε αναπτυσσόμενε χώρε άλλαξαν σημαντικά. Ε, είχαμε μια σημαντική συζήτηση, α πούμε, λίγο πριν για την Κίνα, την Ιδία, τη Βραζιλία που εποφελήθηκαν τα τελευταία χρόνια και εποφελούνται από την παγκοσμιοποίηση, την παγκόσμια αγορά αλλά όλες ε, καθυστέρησαν και υπάρχει κίνδυνος να τεθούν στο περιθώριο τι προτείνει η Επιτροπή για να μην υπάρξει χάσμα ανάμεσα στους δύο, να δοθεί περισσότερο ενδιαφέρον και μέσα στις ε, αργοπορημένες ε, και χρειάζονται βέβαια και δικές τους μεταρρυθμίσεις εσωτερικές ε, και η άποψη της κυρία Σαϊφή δείχνει καθαρά αυτές τις απόψεις της Επιτροπής ε, εμπλουτίζει γιατί, γιατί προτείνει διάφορες πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την εστίαση αυτής της Επιτροπής εξηγήσαμε μερικά πράγματα και την υποστήριξη επίσης λοιπόν στην άποψη της κυρία Σαϊφή και στην ομάδα μου θα προτείνουμε διάφορες τροπολογίες ε, για ένα καλύτερο συντονισμό όλων αυτών των σχεδίων, ε, των επιχειρήσεων ε, και για τους ανθρώπινους πόρους όπως ανέφερε ο, προ... ο εκπρόσωπος του ΟΣΑ και ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε την ένταξη στην παγκόσμια αγορά με μια διευκόλυση της ένταξης της περιφερειακής. Έτσι ε, θα βοηθήσουμε και τις δύο πτυχές και είναι αυτά κεντρικά σημεία λόγω των θετικών αποτελεσμάτων στη μάχη κατά της στόχιας. Ευχαριστώ, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Από τους Ευχαριστώ. Είναι τεράστια ευκαιρία που προσφέρεται και στις δύο. Επιτροπές να δούμε πώς από την ε, βοήθεια, να περνάμε σε εμπορικές συναλλαγές. Ίσως λοιπόν θα ήταν καλό να μειωθεί σε το χρόνο η ανάγκη για αναπτυξιακή βοήθεια, ώστε να αναπτυχθούν οι σχέσεις εκείνες που θα μας οδηγήσουν σε εμπορικές συναλλαγές. Και έτσι ρωτώ, γιατί προσφέρουμε βοήθεια για να εξασφαλίσουμε την ε, ασφάλεια και την ησυχία μας στην Ευρώπη. Γιατί μας τύπτει τη συνείδησή μας που δεν αντέχουμε πια να βλέπουμε τα παιδιά που λιμοκτονούν στην Αφρική. Και πάντως, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι όταν περνάμε συνθήκες εμπορικών συναλλαγών αλλάζουν οι όροι και μιλάμε όχι πλέον συγκινησιακά, αλλά με αντικειμενικό τρόπο, με ουδέτερο τρόπο. Ξέρουμε ότι για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Και είναι δύσκολο και για μας συνδυσιακά να το αντέξουμε, αλλά και να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ σε ποιον δίνουμε την αναπτυξιακή βοήθεια, σε ποιον αν προσφέρουμε εμπορικές συναλλαγές. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με κράτη και αρχές με τις οποίες μπορούμε να συναλλαγόμεθα, αλλά ο άκληρος αγρότης πάλι παραμένει ε, αβοήθητος πολύ συχνά. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ αναπτυξιακή βοήθεια και εμπορικών συναλλαγών. Θα θέλω να δω τη δική σα ε, ματιά σε αυτό το πράγμα. Γιατί εάν ε, από τη σκοπιά με κυβερνητική οργάνωση που δουλεύει στι χώρε αυτέ και προσπαθεί να βοηθήσει για να δώσει τι δυνατότητε στους ε, πολίτες των φτωχών αυτών κρατών να σταθούν τα πόδια του, πάλι χρειάζονται χρήματα. Άρα πάλι, πάλι τα πράγματα ξαναγυρνάνε στην αρχή, στην αφετηρία. Ίσως όμως και να μην είναι τόσο σωστή η απλούστευση. Εγώ λοιπόν έχω συμμετάσχει στην ΑΚΕ, στην κοινοβουλευτική συνέλευση, και με φορές, μερικές φορές με δυσφορία διαπιστώνω ότι οι κανόνες μας οι εμπορικοί εμποδίζουν την ανάπτυξη των κρατών. Γιατί μπορεί για τις πρώτες ύλε να μην έχουμε τελωνιακούς δασμούς, αλλά επιβάλλουμε τελωνιακούς δασμούς για την εισαγωγή ε, καφέ, σοκολάτας και το καθεξής και ως εκ τούτου ή ε, κατεργασμένων προϊόντων. Και έτσι προχωρούμε με τη συμπεριφορά αυτή, εμποδίζοντας τις χώρες αυτές να σταθούν στα πόδια τους, να αναπτύξουν τη δική τους τη βιομηχανία. Και αυτό βέβαια με, μια, με ε, δεδομένου τον κίνδυνο για τις εγχώριες ευρωπαϊκές δηλαδή, θέσεις εργασίας. Άρα είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία αυτή την οποία θα πρέπει να εξασφαλίσουμε, αλλά πρέπει να την κοιτάξουμε. Τώρα μαθαίνω ότι η Μποτσουάνα έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης αδαμαντοκοπτών. Και είναι πολύ λογικό το να μπορεί μια χώρα η οποία έχει εξόρυξη αδάμαντος να μπορεί και να ε, το κατεργάζεται το προϊόν αυτό και να μην το εξάγει μόνο ως ε, ακαταργαστή πρωτήλη. Άρα θα πρέπει να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε και ως προς τη φορολογία και ως προς τη δημοκρατία, γιατί διαφορετικά θα μπορέσουμε να έχουμε ποτέ ισότιμες εμπορικές σχέσεις με τις χώρες αυτές. Και μια άλλη παρατηρήση. Πράσινη ανάπτυξη. Αϊφόρο πράσινη ανάπτυξη, η οποία είναι προ όφελο των αυτών, αλλά ολόκληρου του πλανήτη. Γύρω από αυτήν πρέπει να περιστραφεί οτιδήποτε πράξουμε, συμπεριλαμβανομένη και τη διαφάνεια. Μίλησατε για τι προεδρικέ εκλογέ στι ΗΠΑ σήμερα. Ελπίζουμε να μην εκλεγεί ο λάθο υποψήφιο, γιατί έχει υποσχεθεί ότι θα καταργήσει την νομοθεσία του Fines και αυτό θα έχει καταστροφικέ συνέπειε για τι ε, χώρε του τρίτου κόσμου. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την παρουσία σα εδώ και βέβαια όταν έρθει η ώρα θα καταθέσω πετροπολογίες. Ευχαριστώ κυρία Κέλλερ εκ μέρου των Πρασίνων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την έκθεση. Έχω κάποιες ερωτήσει για τον κύριο Ταλγού του ΩΣΑ και ξεκινώντα, ίσως κάτι να μην άκουσα καλά αλλά λέτε ότι ο ΣΑ εξετάζει το πώς μπορούν οι επενδύσεις μας να βοηθήσουν στην ανάπτυξη. Έτσι δεν είναι. Από την άλλη όμως δεν κατάλαβα πώς αυτά που κάνετε βοηθούν στην ανάπτυξη. Εσείς λέτε ότι βοηθάτε στις επενδύσεις, αλλά ε, από τις επενδύσεις στην ανάπτυξη πώς φτάνουμε. Πώς βοηθάτε τις επενδύσεις να βοηθήσουν την ανάπτυξη. Και αυτό το λέω γιατί και εσείς ε, χρησιμοποιείτε τον όρο επενδύσεις συνέχεια. Πρέπει δεν να πω ότι η συνθήκη της Λισαβόνας δεν μιλάει πιθανά για επενδύσεις, για ανάπτυξη μιλάει. Για αναπτυξιακούς στόχους μιλάει. Για κατάρριξη της φτώχειας μιλάει. Η εκρίζωση της φτώχειας. Και άρα ερωτώ, εάν το PCI στρέφεται κατά του PCG ή εάν σκοπεύεται να ενσωματώσετε τα θέματα αυτά στις προτάσεις σας. Μπορούμε να μιλούμε για αναπτυξιακούς στόχους ή όχι. Επίσης, πάνω σε ποιον ορισμό της ανάπτυξης στηρίζεστε στο έργο σας. Ε, επίσης, Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες περαιτέρω για τις επενδύσεις είτε άμεσε επενδύσει χαρτοφυλακίου, παραγωγικέ επενδύσει ή ό,τι άλλε επενδύσει υπάρχουν για την Αφρική συγκεκριμένα. Τι, τι επενδύσει μπορούμε να βρούμε στην Αφρική, εάν υπάρχουν δεδομένα. Επίσης για σας, ποιε είναι οι ελάχιστες προδιαγραφές για τις ε, επενδύσεις εκείνες οι οποίες θα βοηθήσουν, θα υποβοηθήσουν την ανάπτυξη και τι μέτρα προτείνετε. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις μου για την έκθεση δε. Θα ήθελα να πω ότι συμμεριζόμαστε πολλές παρατηρήσεις της συγκήτριας. Είναι πολύ σημαντικό το ότι υπογραμμίζεται το ότι το εμπόριο και οι επενδύσεις δεν είναι πάντοτε ισόφελος της ανάπτυξης, δεν είναι αυτός σκοπός και ότι πρέπει να προωθηθούν κατά τρόπο ώστε να στηρίξουν την ανάπτυξη, γιατί δεν το κάνουν αυτομάτως, δεν στηρίζουν την ανάπτυξη αυτομάτως. Αυτά λοιπόν. Και θα πρέπει να λέμε νομίζω να δείχνουμε τον τρόπο μας πόσο σημαντικό είναι το να έχουμε εταιρικές, εμπορικές σχέσεις θεμητές τόσο όσον αφορά τις περιβαλλοντικές αλλά και τις κοινωνικές ε, προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές και όχι πάση θυσία εμπορικές σχέσεις. Για τις εμπορικές ε, σχέσεις δεν θέλω να πω ότι σπάνια αναπτύσσονται εμπορικές σχέσεις σε ισότιμους όρους Κάποιο εταίρο συνήθω είναι πιο ισχυρό, κάποιο είναι λιγότερο ισχυρό. Και αν δούμε και τις ε, συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές φορέ υπάρχουν χώρες οι οποίε δεν θέλουν να τι προσυπογράψουν, να τι δεχθούν, αλλά υποχρεούνται διότι διαφορετικά κινδυνεύουν όπω απειλούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να χάσουν άλλα πλεονεκτήματα. Άρα δεν βλέπω ακριβώ ποιο είναι το ισότιμο πεδίο ε, συναλλαγής εδώ. Επίσης σημειώνεται ότι θα πρέπει να ενισχύονται και άλλες πολιτικές, φερειπίν γεωργική πολιτική. Αλλά και πάλι σημειώνω ότι ο κύριος στόχος πρέπει να είναι η εκρίζωση της φτώχειας, η ανάπτυξη και όχι ε, η πρόταση λύσεων που ενδεχομένω να ανατρέπουν τους στόχους αυτούς. Δυστυχώ πολλά είναι τα σημεία, είτε στην γεωργική πολιτική, είτε στην αλληλευτική πολιτική, την εμπορική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση που τείνουν προ την αντίθετη προς το αντίθετο αποτέλεσμα. Στην τελευταία μας συνεδρίαση πρέπει να πω ότι πάλι είχαμε διαπιστώσει μια κάποια βαρέσκεια από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. δεν διαδετύπωσε δηλαδή ε, για το δικό της έργο. Δεν ε, σημείωσε την ε, ασυνέπεια και ασυμβατότητα μεταξύ τη πολιτική μα προ τα τρίτα κράτη και της και αλληλευτικής κτλ. πολιτική που επεσήμανα νωρίτερα. Ερωπό λοιπόν τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταλήξει κάποια διαφορετικά ε, συμπεράσματα. Διεπιστώνεται ότι αυτή η στρατηγική έχει βοηθήσει για την πραγματική ανάπτυξη. Μπορούμε να διαπιστώσουμε κάποια βελτίωση. Γιατί μάλλον βελτίωση δεν βλέπουμε, μάλλον οπισθοδρόμηση διαπιστώνεται. Άρα πρέπει να κάνουμε αυτές τις προσπάθειες και να ενισχύσουμε τα σχετικά σημεία. Ευχαριστώ πολύ ο κύριο Σόλτς εκ μέρους της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ. Και θέλω να δώσω κάποιες ε, βασικές τοποθετήσεις για την πρόταση εκθέσεως και για τη διάσταση του ζητήματος. Ξεκινώ ευχαριστώντας την εισηγήτρια, η οποία επισημαίνει ελλείμματα, προβλήματα στην αναπτυξιακή πολιτική, την εμπορική πολιτική, την πολιτική των επενδύσεων. Όπου θέλω να σημειώσω ότι ο διάβολος κρύβεται συνήθως λεπτομέρειες και κατά την περαιτέρω επεξεργασία της εκθέσεως με τις τροπολογίες ακριβώς πιστεύω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε αυτές τις λεπτομέρειες. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν στην Νέα Υόρκη Είχαμε μια διεξοδική συζήτηση με τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, αρμόδιο για θέματα ανάπτυξης. ο οποίος σημειώνει ρητά τα θέματα στα οποία θα πρέπει να στραφούμε και θέλω να τα φέρω εδώ στη συζήτηση και είπε ότι παραμένουν τα 2,5 δισεκατομμύρια ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση σε συνθήκες υγιεινής. Παραμένουν τα ποσοστά των παιδιών που πεθαίνουν κάθε μέρα. Μόνο και μόνο γιατί δεν έχουν τουαλέτα. Να χρησιμοποιήσουν. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε γιατί τι πράγμα ακριβώ συζητούμε. κυρία Κέλλερ επισήμανε ακριβώς αυτό ότι πρέπει να δούμε ποια είναι η ισορροπία μεταξύ αναπτυξιακή βοήθεια, εμπορικών σχέσεων και πώ θα μπορέσουν τα κράτη από το τοπικό, το περιφερειακό, το εθνικό επίπεδο να εξασφαλίσουν εκείνη τη στήριξη που θα τους επιτρέψει να επενδύσουν στην αλλαγή αυτή και αντίστοιχα εμείς από πλευράς μας θα πρέπει να εντοπίσουμε ποια είναι η δική μας ευθύνη και ρωτώ, πέρα από όλες τις μεγάλες αρχές και αξίες, ξέρουμε γιατί πράγμα μιλάμε. Πώς μπορούμε να προσφέρουμε μια τίμια, ανοιχτή, διαφανή συνεργασία με τα κράτη του Νότου. Πώς μπορούμε να προσφέρουμε ευκαιρία για πραγματική αλλαγή των συνθήκων διαβίωσης των ανθρώπων αυτών. Πώς πρέπει να ρυθμίσουμε τον τομέα ή να διαρρυθμίσουμε τον τομέα των υπηρεσιών, της ε, υγείας, κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετήσουμε όχι απαραίτητα με τα δικά μας μέτρα, την αποτελεσματικότητα και την ανάπτυξη, πραγματική ανάπτυξη στα κάτι αυτά. Και άρα έχω να διαρωτήσω γιατί να για την συγκεκριά. Στο κείμενο γίνεται λόγος πολύ για, να... για χρηματοοικονομική βοήθεια στον τομέα των υπηρεσιών που θα πρέπει να προχωρήσει κτλ. Και θέλω να ρωτήσω οι κρατικές επενδύσεις σε σχέση με τις ιδιωτικές επενδύσεις, σε τι σχέση βρίσκονται πρόσθετα χρηματοοικονομικά μέσα προτείνονται για να οργανωθεί και να εμπλουτιστεί, θα έλεγα, αυτή η πολιτική των επενδύσεων και περιλαμβάνονται σε αυτά τα επιπλέον κονδύλια, σε αυτή την πρόταση, τόσο κρατικά όσο και ιδιωτικά κεφάλαια. Θα κινητοποιηθούν δηλαδή αυτά τα κεφάλαια. Και επίσης, Εάν ένα, εάν ένα φορέας ε, θελήσει να χρηματοδοτήσει αυτό που λέγαμε τώρα, δηλαδή την αποχέτευση, συνθήκες υγιεινής, τουαλέτες κτλ. για τα κράτη αυτά. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα κριτήριο με βάση το οποίο θα προσφέρουν η δημόσια αλλά και η ιδιωτική πλευρά, η επενδυσιακή, μια πραγματική βοήθεια για τα κράτη αυτά. Γιατί βλέπουμε ότι ε, όπως έγινε παραδείγμα τη συζήτηση με τον φόρο για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές είναι αρκετά περιορισμένες οι πραγματικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσει και άρα θα πρέπει να είμαστε πιο επιφυλακτική ενδεχομένω και πιο προσεκτική και να κοιτάξουμε πολύ μεγαλύτερη προσοχή και συγκεκριμένα τις προτάσεις που διατυπώνονται μέσα στην έκθεση για να έχουμε πιο μεγάλα απτά, συγκεκριμένα και διαφανή αποτελέσματα. Merci. Σας ευχαριστώ. Να υπενθυμίσω ότι για την έκθεση αυτή θα πραγματοποιηθούν και άλλες συζητήσεις. Ε, δεν είναι η οριστική, η τελική. Μήπως ε, Κάτι θα ήθελε να πει η Επιτροπή και ο Ντενί Μπαρέσ. Αλλά παρακαλώ σύντομα αν λάβετε το λόγο γιατί δεν έχουμε και τόσο χρόνο για να φέρουμε σε πέρα στη μέση διάταξή μας. Αλλά κάτι θέλετε να πείτε. Ευχαριστώ. Πολλά έχω να πω και υπήρξαν και πολλές παρεμβάσεις αλλά θα είμαι σύντομος. Τέλος πάντων θα προσπαθήσω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έγγραφο εργασίας. Ε, συμφωνούμε με τη γενική ιδέα και υπάρχουν και πολλά σημεία σύγκλησης με τη δική μας ανακοίνωση. Θα ήθελα να υπενθυμίσω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα είναι ένα τεράστιο εγχειρίσμα μεταξύ της Επιτροπής Εμπορίου και τη Επιτροπής ανάπτυξη. Ε, είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα ε, ανάπτυξης πολιτικής, ενδεχομένως το βέλτιστο παράδειγμα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και η ιδέα αυτής της ανακοίνωση, κάτι ακόμη που θα ήθελα να πω, δεν ήταν να αλλάξουμε την πολιτική μας απλώς για να την αλλάξουμε, απλώς για να προστα... προσαρμοστούμε ε, στην... Ε, κατάσταση που είναι η ανάδυση νέων οικονομιών, ε, κάτι το οποίο βέβαια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και στη δική μας ευθύνη. Είναι κάτι το οποίο αναφέρεται και στο δικό μας ε, έγγραφο και στο έγγραφο της ε, εισηγήτριας. Μερικά πράγματα που θα ήθελα να τονίσω είναι τα εξής για το έγγραφο εργασίας τουλάχιστον. Είναι καταρχάς η σημασία της βοήθειας για το εμπόριο και της σημασίας για την καταπολέμηση της φτώχειας και την ανάπτυξη των χωρών. Αυτό το, το οποίο θα έπρεπε να είναι κυρίαρχο είναι ο ρόλος των ε, εσωτερικών πολιτικών και της πλήρους ε, εξοικείωσης των χωρών αυτών, ε, γιατί αυτές βρίσκονται στη θέση του οδηγού και μόνο εκείνες μπορούν να τα καταφέρουν. Εμείς μπορούμε απλώς να τις βοηθήσουμε, να τις βοηθήσουμε, να τους διευκολύνουμε στις εσωτερικές τους πολιτικές. Όσον αφορά τώρα η εμπορική βοήθεια και το στόχο αυτό, πολύ σημαντικό είναι και αυτό, αλλά υπάρχει και το θέμα της κυριότητας που ανέφερα προηγουμένως. Οι χώρες εκείνες πρέπει να αποφασίσουν κατά πόσο πρέπει να, να λάβουν αυτή τη βοήθεια για το εμπόριο και μετά πώς θα τη χρησιμοποιήσουν. Αυτό το, το θέμα της ε, του καλύτερου συντονισμού μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων δωρητών... Ε, είναι εδώ και όσα, όπως είπα, είναι, είναι, είναι πάρα πολύ καλό ε, παράδειγμα καλής συνεργασίας ε, αυτή η περίπτωση. Όμως υπάρχουν και άλλες πτυχές οι οποίες υπερβαίνουν τις καθαρά εμπορικές. Υπάρχει το θέμα ε, ε, υπάρχουν πτυχές που είναι θέμα της ε, Επιτροπής Ανάπτυξης Αναπτυξιακής Πολιτικής, κάτι το οποίο επίσης πιστεύω ότι πρέπει να αναφέρεται στο, κάτι το οποίο επίσης αναφέρεται στο έγγραφο εργασίας. η ανακοίνωσή μα ε, δεν είχε σκοπό να αλλάξει τα πράγματα απλώ για να τα αλλάξει, αλλά για να βελτιώσει την κατάσταση. Αν δει κανεί τα μέσα που υπάρχουν, ε, εξελίσσονται συνεχώ. Υπάρχει το νέο σύστημα γενοτιευμένων προ... προτιμήσεων, υπάρχουν νέε συμφωνίε με τι ε, χώρε που συμπεριλαμβάνουν διάφορε πτυχέ, όπω ε, τι συνθήκε εργασία, το περιβάλλον, τι επενδύσει. Έχουν, έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ αυτά τα μέσα. Υπάρχει το θέμα της ε, περιφερειακής εμπορικής ε, ολοκλήρωσης. Είναι γεγονός, ε, είναι αρκετά έντονο το έγγραφο εργασίας προς αυτό. Αν το θέμα αυτό αφορά τις εμπορικές συμφωνίες, πιστεύουμε ότι η δική μας προσέγγιση αποφέρει καρπούς. Ένα κατάλογο τώρα δράσεων που συμπεριλαμβάνεται στο έγγραφο εργασία, θα ήθελα να το σχολιάσω και αυτό. Αν δει κανεί τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει τη βοήθεια για το εμπόριο, όλα αυτά τα ζητήματα καλύπτονται ήδη. Είτε πρόκειται για ε, για τις υποδομές ή για άλλου είδους ε, ε, ανάπτυξη ικανοτήτων. Είναι όμως οι εταίροι μας αυτοί που σε τελική ανάλυση αποφασίζουν εάν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα που λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το εμπόριο για κάτι άλλο και αν ε, για το εμπόριο, για αν το χρησιμοποιήσουν, τα χρησιμοποιήσουν για το εμπόριο, πώς θα τα χρησιμοποιήσουν. Αυτά. Να σταματήσω εδώ. Euh, σας ευχαριστώ ναι, Για ένα λεπτό μόνο. Μόνο για λόγους αυρότητας, γιατί έχουμε καθυστερήσει πολύ ένα λεπτό, όπως έχουν συνηθίσει οι βουλευτές να μιλάνε στην Ολομέλεια. Αν έχετε κάτι σημαντικό λοιπόν να πείτε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Καταρχά, υπόθηκε βεβαίω ότι δεν μπορεί η ανάπτυξη η μόνη τη να λύσει κάθε πρόβλημα. 40 δις βοήθειας λαμβάνει η Αφρική πολύ περισσότερο καταναλογία να πω ότι η Ινδία που έχει περίπου ένα δισεκατομμύριο κατοίκους. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ε, προωθήσουμε αυτούς τους πόρους με καινοτόμα μέσα επενδυσιακά ταμεία κτλ. Και το πιο σημαντικό, να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να ενισχύσουν την τους, ε, το αναπτυξιακό του δυναμικό. Και βέβαια αυτό δεν αναφέρεται μόνο στην σχέση μεταξύ εμπορικών σχέσεων και ανάπτυξη. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να αναπτύξουμε, μπορούμε να ενισχύσουμε την ανάπτυξη με τι εμπορικέ σχέσει και πάνω απ' όλα να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές για καλές πολιτικές, για να προσδιορίσουν τις ικανότητες τους, τις προτεραιότητες τους, το πλαίσιο πολιτικής τους. Και πολύ σημαντικό είναι να δείξουμε ότι μπορούν να έχουν κανόνες λειτουργίας για τι επιχειρήσει και βέβαια μπορεί να κοιτάξουμε εν τέλει και πολύ σημαντικού τομεί όπω αυτών τη γεωργία, τη εξωτερική βιομηχανία. και να ενθαρρύνουμε επενδυτέ, αλλά και κοινωνίε ολόκληρε για εμπορικές σχέσεις στον Ευχαριστώ εκ μέρου ε, της συγκεκριτή, ο κύριος Δαβίτ. Ευχαριστώ σύντομα. Να ευχαριστώ του συναδέλφους που πήραν το λόγο και την Επιτροπή και τον κύριο Καρίμ Ντεού βέβαια και σίγουρα θα μεταβιβάσω στην κυρία Σάιφη αυτή μάλλον θετική προσέγγιση όλων των ομάδων και θα περιμένει και τη συνεισφορά όλων των συναδέλφων στην έκθεση της. Ευχαριστώ. Ναι. Και εμείς περιμένουμε την έκθεση αυτή για την επόμενη συνάντηση στο τέλος του Νοεμβρίου. Και τώρα ερχόμαστε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης έχει πολλά. Συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και της Κολομβίας και του Περού αφετέρου. Πρόκειται για σημαντική συζήτηση εδώ στο Κοινοβούλιο. Έχουμε δύο ταυτόσιμες τροπολογίες που κατατέθηκαν που απορρίπτουν τη συμφωνία. Και θέλουμε τον Ιούνιο του 2012 ψήφισμα του Κοινοβουλίου να το ακολουθήσουμε που ζητούσε από την Κολομβία και το Περού να έχουν ένα οδικό χάρτη για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος και των κοινωνικών παρομοίων και Είχαμε μια συζήτηση με μια κείμενα τις δύο χώρες και χαιρόμαστε που τον κύριο Ροντρίγκο Ριβέρα Σαλαζάρον, πρέσβη της ε, Κολομβίας και τον κύριο Τσάβης από ε, που είναι υπουργό επί του πρωτοκόλου και του Περού. Έχετε το λόγο και για να σεβαστούμε και τα κοινωνικά δικαιώματα των διερμηνέων μας. Έχουμε οκτώ λεπτά για κάθε παρέμβαση για τους δύο εκπροσώπους των χωρών. Μήπως μπορείτε να τα σεβαστείτε αυτά. Μια σύντομη συζήτηση πριν από το διάλειμμα για το γεύμα. Εσείς τα είπατε αυτά, είναι πολύ ογκώδες το θέμα αυτό με και ο δικός μου όγκος, εντάξει, γι' αυτό, <laughs> για, σε αυτό να επίσης αναφέρομαι. Και θα συνεχίσω αγγλικά. Αγγλικά θα συνεχίσω λοιπόν. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι σε σχέση με αυτά που έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια για τις εμπορικές συμφωνίες. Είναι η πρώτη φορά, εξ όσων γνωρίζω, ότι ε, για πρώτη φορά κυρίαρχα κράτη αντιμετώπισαν το θέμα με έναν πάρα πολύ θετικό τρόπο, ανταποκρίθηκαν με πολύ θετικό τρόπο στο αίτημα που κάναμε πριν από ε, πέντε μήνες. Ε, δεν γελιοποιηθήκαμε προσπαθώντας να επιβάλλουμε κανόνες σε νόμους σε άλλες χώρες, σε χώρες στις οποίες δεν έχουμε καταφέρει να, επιβάλλει, να επιβάλλουμε στις δικές μας χώρες, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευτυχώς δεν συνέβη κάτι τέτοιο και δεν ήμασταν κακοί ενώπιον χωρών που αποφάσισαν να είναι εταίροι μας. Ε, ζούμε σε έναν ε, κόσμο που ευημερεί και ε, θα ήθελα να επικροτήσω τις, την κυβέρνηση της Κολομβίας και του Περού. Ε, κάθε μέρα θέλουμε να επιτυγχάνουμε έναν καλύτερο κόσμο για το μέλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις συζητητές και τους ε, που με βοήθησαν, ε, τον Μπέρντ Λάγκε για την προηγούμε, το προηγούμενο ψήφισμα, το οποίο είχε βασιστεί στην καλή πίστη ε, και την αλλαγή της προσέγγισης που όπως ε, είχαμε προγραμματίσει ε, εστέφθηκε με επιτυχία. Όπω φαίνεται άλλωστε και από τα έγγραφα που λάβαμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τι κυβερνήσει των δύο χωρών. Ε, τους ε, πρέσβεις τους ε, και το προσωπικό και των δύο πρεσβειών. Ε, συνεργαστήκαμε πάρα πολύ και θα ήθελα να διαβιβάσετε και τις ευχαριστίες μας στους προκατόχους σας με τους οποίους ξεκινήσαμε την όλη διαδικασία. Τούτων λεχθέντων ε, θα ήθελα να επικεντρωθώ τώρα στο έγγραφο, να σας υπενθυμίσω μία ακόμη φορά ότι μιλάμε για δημοκρατικές κυρίαρχες χώρες οι οποίες ε, θελήσαν, ε, θελήσαν να ανταποκριθούν θετικά στο, στην έκκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καλύτερη επι, επι, περιβαλλοντική προστασία, καλύτερη εποπτεία της κοινωνίας των πολιτών. ανταποκρίθηκαν λοιπόν σε σχέση σχέση με αυτούς τους στόχους. Ε, στα έγγραφα που έστειλαν οι προσβίες φαίνεται ότι είναι ε, ότι δεσμεύονται οι χώρες αυτές για τους στόχους αυτούς, ε, τα οποία βέβαια ανταποκρίνονται πλήρως στον, στην έκκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα κληροδότημα που οι κυβερνήσεις θα αφήσουν στις χώρες τους. Είμαι βέβαιος ότι οι μελλοντικές γενναίες δεν θα το ξεχάσουν. Δεν μπορούμε να ξεχνούμε επίση και αυτά είναι τα δύο συμπερασματικά μου σχόλια, ότι η εμπορική συμφωνία μεταξύ Κολομβίας και Ηνωμένων Πολιτειών ισχύει ήδη και ότι τον Ιούνιο το ψήφισμά μας πρό, ε, πρότεινε, πρότεινε την οργάνωση μιας ακρόασης σε μία από τις ε, πρωτεύουσε ε, των Άνδεων ε, κατά του ερχόμενου μήνε και θα αποσταλεί σχετική, έργο ε, και στην Επιτροπή ε, Διεθνούς Εμπορίου αλλά και στην Επιτροπή ε, Νομικών Υποθέσεων. Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε πλέον την υποστήριξή σας ε, για το ψήφισμα αυτό, το οποίο μπορούμε πιστεύω να, ψηφίσουμε, να υπερψηφίσουμε στην επόμενή μας ε, ε, συνεδρίαση, γιατί οι βασικές μας αξίες την χάνουν πλήρου σεβασμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. η αυτού εξοχότη του κυρίου Σαλάζα θα παρουσιάσει τον οδικό χάρτη της Κολομβίας. Gracias, eh, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να σε ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου προσφέρετε να προσθέσω προφορικά τα όσα ήδη σε μια επιστολή στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχα απευθύνει της 26 Οκτωβρίου. Εξ ονόματος της κυβέρνησης της Κολομβίας και τις σκέψεις μας για το ψήφισμα το πολιτικό της 13 Ιουνίου φέτος από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκεί αναγνωρίζεται ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στα ανθρώπινα δικαιώματα, στα εργασιακά, περιβαλλοντικά, στην Κολομβία και στο Περού Ταυτόχρονα όμως εκφράζονται μερικές ανησυχίες για θέματα που υπάρχουν πάντα, που εκκρεμούν και στο ψήφισμα αυτό το πολιτικό που ε, προτείνει μια, ένα οδικό χάρτη διάφανο για να βελτιωθεί η γενική κατάσταση και στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα εργασιακά και μια υφόρο ανάπτυξη όλα αυτά που έχουν σχέση με το διμερές εμπόριο και με το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση της Κολομβίας απεφάσισε μετά την επίσκεψη του Μάριο Νταβίδε και Βερλάγκε στην Μπογκοτά μετά την επίσκεψη στον πρόεδρο Σάντος και την ε, Βουλή αποφάσισε σε ανώτατο επίπεδο μια, προχωρήσει τη σύσταση μιας ομάδος ε, δια, ε, ώστε τα θέματα αυτά να αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης ε, και να αναφέρουν τα όσα έκανε η Κολομβία μέχρι τώρα αυτό ακριβώς πραγματοποιήσαμε για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις ε, και στα ανθρώπινα τα εργασιακά, τα περιβαλλοντικά και τι θα κάνουμε τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια και να συμπληρώσουμε τη σχετική πληροφορία με διάφορες ανακοινώσεις που έχουν άμεση σχέση με την εμπορική συμφωνία. Γι' αυτό ακριβώς ε, στην επιστολή της 26 Οκτωβρίου στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχαμε την ευκαιρία να πούμε ότι πέρα από δικό χάρτη έχουμε και ένα πραγματικό πρόγραμμα δράσης ε, που είναι δεσμευτικό και που θεσμικά με νόμο υιοθετήθηκε μια ανάπτυξης ε, με τους στόχους, ε, τις στρατηγικές, τις προτεραιότητες της κυβερνησής μας υπό τον πρόεδρο Σάντος από το 2010-2014 σχέδιο που υιοθετήθηκε από την ε, νομοθετική μας εξουσία, την ε, Βουλή μας μετά από πολλή δουλειά και με την επεξεργασία και την... Ε, και συμμετείχε επίσης η κοινωνία των πολιτών μέσω σχεδίων προγραμματισμού και επίσης με τις ε, διάφορες εθνοτικές μειοψηφίες ε, τα συζητήσαμε αυτά γιατί ίσως υπήρχαν και σημαντικές αποφάσεις που θα τους επηρέαζαν, θα τις επηρέαζαν. Και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στείλαμε την επιστολή αυτή μαζί με μια προσεκτική απαρίθμηση των μέτρων των συγκεκριμένων μέτρων και τους συγκεκριμένους στόχους, σε τι προχωρήσαμε σε αυτά τα θέματα, ανθρώπινα δικαιώματα, εργασιακά, περιβαλλοντικά, τι ακριβώς υιοθετήσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια στην Κολομβία. Είναι 56 μέτρα συγκεκριμένα, σαφή, ρεαλιστικά, φιλόδοξα και εφαρμόσιμα, πραγματοποιήσιμα που δείχνουν τις φιλοδοξίες, τους στόχους της Κολομβίας ε, στους τομείς αυτούς και έτσι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μπορούσε να ασκήσει ένα έλεγχο, μια παρακολούθηση, μια εποπτεία για το πώς όλα αυτά πραγματοποιούνται από τα διάφορα Υπουργεία και από τις αρχές που συμμετέχουν στην ε, υλοποίηση όλων αυτών και επίσης 100, παράγουν από 100 ειδικά μέτρα για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους και με 36 συγκεκριμένα, συγκεκριμένους τομείς ε, όπου σημειώθηκε βελτίωση. Επίσης ένα παράρτημα στην επιστολή με την σημαντική πρόοδο μετά από τα συγκεκριμένα αυτά μέτρα και τα τους τρεις-τέσσερις τελευταίους μήνες και εμείς στη χώρα μου διατηρούμε αυτό το ρυθμό με μέτρα κατάλληλα συγκεκριμένα για τους τομείς αυτούς και την πρόθεσή τους και την υλοποίησή τους. Περιλαμβάνουν τα μέτρα αυτά διάφορους τομείς ε, με προγράμματα στρατηγικής 12 μέτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επίσης ενίσχυση της δικαιοσύνης ένα μέτρο, προστασία ατόμων σε κίνδυνο 5 μέτρα, ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, και με διάφορους φορείς, 4 συγκεκριμένα μέτρα, κατά της αντιμορρησίας φόρος, ε, νόμους τέσσερα μέτρα, βελτίωση του διεθνούς διαλόγου κυρίως με την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω σε αυτό το τομέα, δύο μέτρα και επίσης 13 ειδικά αποτελέσματα που έχουμε προχωρήσει στα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουν σχέση με τους στόχους αυτούς και τα μέτρα αυτά. Όσον αφορά το περιβάλλον, την ανηφόρα ανάπτυξη, Εκεί προχωρήσαμε σε μια ταξινόμηση των μέτρων. Το πρώτο από αυτά είναι η Κολομβία που τέθηκε επικεφαλής του Ρίο συν 20 για μια υφόρα ανάπτυξη στην συνάντηση αυτή και επίσης ε, την πραγματοποίηση με την εφαρμογή μέτρων 11 μέτρα για τα δάση, εφαρμογή για την βιοπικιλότητα 5 μέτρα και εφαρμογή πραγματική των προδιαγραφών όσον αφορά το είδωρ 12 μέτρα και εφαρμογή όσον αφορά την εξόριξη φυσικών πόρων 10 μέτρα και εκτό ε, θελοντική εργασία όσον αφορά το περιβάλλον και εφόρο ανάπτυξη με 4 μέτρα. Έβδομο, ενίσχυση του κοινωνικού διάλογου σε θέματα εφοροανάπτυξης ανάπτυξης κοινωνικού διαλόγου με είναι 8 τα μέτρα 8 κατά τις ατιμορρησίας και στο περιβάλλον 3 ε, μέτρα και ένα το βελτίωση της ε, συνεργασίας για την φόρα ανάπτυξη για το περιβάλλον ε, δύο μέτρα κυρίως με την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης τα συγκεκριμένα πράγματα που πετύχαμε για την φόρο ανάπτυξη με 15 σημεία στα οποία συγκεκριμένα προχωρήσαμε. Το ίδιο κάναμε και όσον αφορά το εργασιακό δικαίωμα με διάφορα μέτρα για να εφαρμοστούν όλα αυτά, μέτρα κατά της ατιμορρησίας, ενίσχυση του κοινωνικού διολόγου... και επίσης με τα διάφορα συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά στις εργασιακές σχέσεις. Πέρα από αυτό, που αποστήλαμε στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα να προσθέσω ότι η ίδια η συμφωνία βοήθησε πολύ πάνω σε αυτά με διάφορες ρήτρε, ε, όλα αυτά που θα σεβαστεί η Κολομβία και από τη στιγμή που η εμπορική συμφωνία θα εφαρμοστεί, θα υιοθετηθεί, η κυβέρνησή μας θα ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή της αιφόρου ανάπτυξης για τον τρόπο με τον οποίο προχωράει η Κολομβία σύμφωνα με το ΑΚΑΤ με το άρθρο για μια καλύτερη διαφάνεια και συμμετοχή του Δημοσίου και το Υπουργείο Βιομηχανίας Τουρισμού θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτό, με την εφαρμογή των αυτών και θα ενισχύσουμε τις δυνατότητες των ε, θεσμικών μας οργάνων για να έχουμε ε, καλύτερη κατάλληλη ανάπτυξη όπως προτείνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο μεγαλύτερο όγκο συνεργασίας ώστε όλα αυτά τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί για την εφόρα ανάπτυξη για το εμπόριο να βοηθηθούν και θα ελέγξουμε ε, θα βοηθήσουμε την ανάπτυξη μέσω συμμετοχής μας και επίσης ε, για την εφόρα ανάπτυξη θα έχουμε συμμετοχή μας με την οργανωμένη κοινωνία και πάνω σε σχετικούς τομείς για την εφόρα ανάπτυξη, το εμπόριο όπως είπαμε και επίσης ένα εθνικό μηχανισμό διαβούλευσης και θεωρούμε ότι θα πρέπει η μόνιμη επιτροπή ε, ελέγχου θα πρέπει, η δικιά μας θα πρέπει να έχουν, να έχει ε, να έχει σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της συμφωνίας την αρμοδιότητα με συμμετοχή επιχειρηματιών, συνδικάτων, ε, εθνοτικών ομάδων, ε, κυβερνητικών και λοιπά και όλα αυτά που δείχνουν ότι πραγματικά συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών. Θα ολοκληρώσω εδώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα σαν αγγείλω ότι παρόλο που δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας της εμπορικής η κυβέρνηση της Κολομβίας θα προχωρήσει τη σύσταση μιας τεχνικής ομάδας για, γενικά για τα ανθρώπινα δικαιώματα τις εμπορικές συμφωνίες στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου με μια εποπτεία κατάλληλο μηχανισμό για τα όσα έχουμε προσυπογράψει εμείς η Κολομβία και με συμμετοχή της οργανωσμένης κοινωνία των πολιτών. Επίσης θα δούμε την φορολογικά και θα Επαναλαμβάνομαι με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των συνδικάτων κλπ. και με το κατάλληλο ποινικό σύστημα για να δούμε την παραβίαση ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και που κανείς θα μπορούσε να απευθύνει παράπονα. Επίσης ενισχύουμε τον πολιτικό διάλογο πάνω σε αυτά τα θέματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. της 19 Σεπτέμβρη μας πέρασε είχαμε νέους όρους αναφοράς στον διάλογό μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από τη στιγμή που θα ισχύσει η εμπορική συμφωνία θα μπορούν να παρακολουθούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν σχέση με την διμερή αυτή εμπορική συμφωνία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ριβέρα. Ο κύριος Αβεστσαβούρα για, από το, για το Περού. Θα είμαι λίγο πιο αυστηρός ε, για το χρόνο, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τη συζήτηση για τα έγγραφα που μας παρουσιάζετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν να ξεκινήσω την παρουσίασή μου, θα ήθελα εδώ στα αξιότιμα μέλη να ζητήσω συγγνώμη για την κυρία Φραγκίλιο, την πρέσβη μας ε, η οποία είναι στο Λουξεμβούργο αυτή τη στιγμή που παρουσιάζει τα διαπιστευτήριά της σαν πρέσβης του Περού και δυστυχώς συνέπεσαν οι δύο ημερομηνίες ε, γιατί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Στρασβούργο στις 13 Ιουνίου τα είχαμε πει όλα αυτά και δυστυχώς ε, δεν μπορέσαμε να αποφύγουμε το να συμπέσουν οι δύο μερομηνίε. Όπως ε, είπε και ο, ο πρόεδρός μας, ε, η κυβέρνηση του Περού είναι υπέρ της παγίω δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, την συμπερίπτωση την κοινωνική, την προστασία του ευάλωτου πληθυσμού, την προστασία του περιβάλλοντος και θα πρέπει ο πληθυσμός να έχει καλύτερο επίπεδο ζωής. Η εμπορική συμφωνία λοιπόν στα πλαίσια αυτά που υπέγραψαν η Κολομβία και το Περού με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και όθηση για την ανάπτυξη αυτή από όλες, τις, από πλευρές είναι ένα εργαλείο που θα μας προσφέρει ανάπτυξη και με τον κατάλληλη σχέση ανάμεσα στο εμπόριο και στην αηφόρο ανάπτυξη. Στα πλαίσια αυτά της συμφωνίας ε, η κυβέρνηση του Περού επεξεργάστηκε ένα κείμενο σχετικά με την εφόρον άπτυξη στο Περού, πανόραμα των θεσμικών οργάνων, πολιτικών, στρατηγικών και στόχων και που το επεξεργάστηκε ε, υπό την εποπτεία Υπουργείου πολά πολλά άτομα, δείχνει τις προσπάθειές μας ε, για να εξασφαλίσουμε την πραγματική προστασία, πρόθεση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών ε, κλπ και όλα αυτά που απασχόλησαν ε, στο ψήφισμά σας στο Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό. Και όλα αυτά βρίσκονται στο Σύνταγμά μας, όπως επίσης και η συμφωνία αυτή η εθνική που ξεκίνησε από το 2002 είναι το σύνολο των πολιτικών, ε, των ε, θεσμικών ε, και με τη συνένεση ανάμεσα στην κυβέρνηση, στις διάφορες πολιτικές δυνάμεις και σε προσώπους της κοινωνίας των πολιτών για να έχουμε πραγματικά μια βάση για την εφόρα ανάπτυξη και να μπορέσουμε έτσι να οργανωθούμε και να προχωρήσουμε δημοκρατικά να τονίσω κύριε Πρόεδρε μερικές πτυχές που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα. Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι σημαντικός πυλώνας της πολιτική μας στο Περού και σε εσωτερικό επίπεδο αλλά και στα πλαίσια της εξωτερικής μας πολιτικής. Είμαστε μέλος και σεβόμαστε τα όσα έχουμε συμφωνήσει στους διάφορα διεθνή φόρουμ όσον αφορά τα ανθρώπινα ε, δικαιώματα και στο φόρουμ το διαμερικανικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Συμφωνία υπό την αιγύδα των ΗΠΑ επίσης ε, προσυπογράψαμε σχετική συμφωνία και θα πρέπει να τονίσω ότι υπήρξε ε, υφυπουργό ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ασχολείται με τα θέματα αυτά, όπως επίσης και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Κοινωνικής Ένταξης πλέον. Και να τονίσω επίσης ότι υπήρξε εθνικό σχέδιο 2012-2016 για την πρόθεση και επίσης ε, αποζημιώσεων στα θύματα παρομοίων διακρίσεων από το 1980 μέχρι το 2000 ε, και επίσης το 2011 υιοθετήθηκε νόμος για την προκαταρκή διαβούλευση με τις ομάδες ε, ε τις μειονοτικές και στα πλαίσια των εργασιακών συμφωνιών και το Μάιο είχαμε το σχετικό νόμο που αποτελεί σημαντική βάση για την προστασία των ε, ομάδων ε, εθνικές μειονότητες μας και όσον αφορά τα εργασιακά θέματα εμείς θέλουμε την ε, το να ξεριζώσουμε τη φτώχεια που είναι βασικές αρχές για την ανάπτυξη της χώρας. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και η υπόσχεση ότι θα στηρίξουμε τα βασικά θαμελιώδη δικαιώματα όπως την συνδικαλιστική ελευθερία, την ε, την δυνατότητα στους συνεταιρίζεστε, όχι καταναγκαστική εργασία και όχι εργασία των παιδιών και σε διεθνέ επίπεδο ε, σε 74 διεθνείς συμφωνίες έχουν προσυπογράψει για να υποστηρίξουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα τα εργασιακά. Επίσης επεξεργαστήκαμε την κοινωνική επιχειρηματική ευθύνη στα πλαίσια του 2011-2013 για την σωστή πρακτική για να μπορέσουν να γίνονται σεβαστά τα όσα έχουν θεσπιστεί εργασιακά και σύμφωνα και με τα όσα έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Εμείς θέλουμε την πρόκληση για μια, ένα ποιοτικό άλμα αυτή η ανάπτυξη να γίνει βάση της ε, κληρονομιάς μας κάθε είδους στη χώρα μας και θέλουμε να προτείνουμε νόμους, ρυθμίσεις, να βοηθήσουμε το περιβάλλον και σαν στόχος για την ανάπτυξη αηφόρο ανάπτυξη, να προστατεύσουμε την υγεία του πληθυσμού μαζί και να προσέξουμε, να φροντίσουμε το περιβάλλον. Θα ήθελα να τονίσω ότι ο πρόεδρος μας τον Αύγουστο παρουσίασε την κρατική πολιτική για το πόσιμο είδωρ και γενικά τα ύδατα και σε αγροτικές περιοχές. Και ιδιαίτερη σημασία έχει ο διάλογος ανάμεσα στο κράτος και στην κοινωνία των πολιτών για μια συμμετοχή πολιτών. Εμείς να λάβουμε υποχρέωση γι' αυτό. Και επίσης ε, θα πρέπει να μπορέσουμε να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν για συνεργασία μεταξύ του κράτους και των κοινωνικών εταίρων βάσει νόμων αποκέντρωσης και το Εθνικό Συμβούλιο Εργασίας και το Εθνικό Συμβούλιο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για την ε, προδιαπραγμάτευση και διάφορες άλλες εθνικές συμφωνίες και την ε, μεχανισμό συμμετοχής ε, στις ε, συμφωνίες του, τις εμπορικές του Περού υπάρχουν ειδικευμένε επιτροπές και στα πλαίσια της συμφωνίας με τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εμπορική συμφωνία να παλάβω την άλλη υποχρέωση από την κυβέρνησή μας ότι από τη στιγμή που θα επικυρωθεί θα ισχύσει στο σύνολό του και κυρίως το άρθρο 9 για να μπορέσουν να συμμετάσχουν όλοι στο Περού στις προσπάθειες αυτές. Και από πολιτικής πλευράς εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε την οικονομία με αποτελέσματα απτά κατά της φτώχειας, κατά της ανισότητας, ε, μείωση της ανεργίας και στα πλαίσια αυτά με την εμπορική συμφωνία έχουμε ένα σημαντικό εργαλείο για την πρόθεση του εμπορίου και μια ποιότητα και στο περιβάλλον, στις κοινωνικές σχέσεις και δυνατότητες επίσης για επενδύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις υπηρεσίες, για τις ανώσιμες πηγές ενέργειας και για το περιβάλλον και για βιομηχανικά βέβαια, βιομηχανικές πτυχές. Εδώ εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο δικό μας Κοινοβούλιο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για τις προσπάθειές σας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανάπτυξη αυτή στα πλαίσια της αμοιβές εμπιστοσύνη και σεβασμού. Και το έγγραφο αυτό δείχνει την προσπάθειά μας και την άνοιξη υποχρέωση και του πληθυσμού μας μέσω πολιτικών και ενεργειών να σεβαστούμε αυτούς τους χαραγμένους στόχους για τα επόμενα χρόνια για να αποφύγουμε προβλήματα και να μπορέσουμε να πετύχουμε την ανηφόρα ανάπτυξη που όλοι μας ε, προσπαθούμε και ευχόμαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δύο λεπτά θα δώσω σε κάθε σκιώδη εισηγητή. Να ζητήσω συγγνώμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο και προτείνω να αφήσω περισσότερο χρόνο στους ε, ε συναδέλφους βουλευτές. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς που θα μας δώσουν 10-15 λεπτά επιπλέον. Κύριος Λάγκη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστώ τις δύο κυβερνήσεις και τους προσβευτές τους εδώ για τις απαντήσεις, ε, για την ανταπόκριση στο ψήφισμά μας που αποτελεί πιστεύω την αφετηρία ενός διαλόγου για νέες σχέσεις με βάση και τις αλλαγές που έχει φέρει, επιφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας ως προς την ισορροπία δυνάμεων, δηλαδή το ρόλο που μπορεί να διδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά βέβαια πιστεύω ότι είναι και προς το συμφέρον της Κολομβίας και του Περού των ιδίων να ενισχύσουν την ανάπτυξή τους. Στο βαθμό αυτό λοιπόν εκφράζω την ικανοποίησή μου γιατί έχουμε εδώ δύο έγγραφα, λεπτομερή, πολύ λεπτομερία για την ε, ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των ανθρωπινών δικαιωμάτων, των προδιαγραφών ε, ασφαλείας των χώρων εργασίας και πρόκειται για πολύ διεξοδική περιγραφή των συνθήκων αλλά και των προοπτικών για το μέλλον. Με ικανοποίηση βλέπω επίσης ότι υπάρχει διαφάνεια σημαντική Μπορούμε να συζητούμε για μέτρα, μπορούμε να συζητούμε δηλαδή για προθέσεις και αυτό δεν είναι αρκεί. Τώρα εδώ έχουμε επί συγκεκριμένα μέτρα, συγκεκριμένα βήματα για το μέλλον και ιδιαίτερος για την κυβέρνηση της Κολομβίας ε, πρέπει να τη συγχαρώ γιατί έχει θέσει το σχέδιό έχει διαθέσει το σχέδιό της στο ίντερνετ και έτσι μπορεί ο καθένας και να το συμβουλευτεί αλλά και να επαληθεύσει ε, τις εξελίξεις, ότι πράγματι δηλαδή ακολουθείται το σχέδιο. Και εδώ ολοκληρώνω λέγοντας ότι πρέπει από κοινού να διαμορφώσουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Έχουμε αποφάσεις από την Επιτροπή για τη θέσπιση μια ομάδα εποπτείας, η οποία και στο μέλλον θα παρακολουθεί τις εξελίξεις μέσα, μέσα από εντατικό διάλογο που πιστεύω ότι μπορεί να συνεχιστεί κατά τρόπο πολύ θετικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πέρμπερ. Ε, Πολύ σύντομα, πρόεδρε. και στο συγγνώμη από το Περού, θα επικεντρωθώ στην Κολομβία, γιατί δεν είχα το χρόνο να μελετήσω το έγγραφο του Περού. Πολύ δουλειά έχει γίνει λοιπόν, πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό και συγχαίρουμε την ομάδα της Κολομβίας για τις προσπάθειές τους και την πρόοδό τους. Πρέπει να πω όμως ότι είμαι κάπως απογοητευμένη. Γιατί λέγεται στον οδικό χάρτη ότι πριν να τεθεί σε εφαρμογή μια συμφωνία εμπορικών συναλλαγών θέλουν συγκεκριμένε προποθέσει να έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Εδώ όμω δεν βλέπω ακριβώ ε, κάτι το συγκεκριμένο στις, ε, στα μέτρα τα οποία εισάγεται όλες αυτές οι οργανώσεις, οι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζι, όλα αυτά γίνανε, έχουν προχωρήσει κατά τρόπο ικανοποιητικό. Εμείς βεβαίως είμαστε ικανοποιημένοι για τις προθέσεις που διαβάζουμε, αλλά πρέπει και να δούμε συγκεκριμένα και αυτά αποτελέσματα. Οι περισσότεροι δικαστές έχουν οδηγήσει ε, σε καλύτερη λειτουργία των ε, δικαστηρίων έχουν οδηγήσει σε αποτελεσματική απονομή δικαιοσύνη. Επίση, είναι πολλέ οι μη κυβερνητικέ οργανώσει που διαμαρτύρονται, πρέπει να πω, γιατί δεν του επιτρέπει η συμμετοχή σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αισθάνονται ότι έχουν αποκλειστεί και κάνουν παρατηρήσεις πίν ε, για προστασία του περιβάλλοντος και άλλα ζητήματα που θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε. Η ε, επιδόση παραδείγματι στον χώρο της εξόρυξης άνθρακα είναι πολύ ε, κακές και θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το σημείο. Βέβαια τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των, των ε, έργων εξόρυξης. Ξέρω ότι δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά ρωτώ επιπλέον τι πρόοδο μπορούμε να σημειώσουμε. Βεβαίως έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος, αλλά χρειάζεται περισσότερη πρόοδος ακόμη και πρέπει να πω ότι αισθάνομαι μια κάποια απογοήτευση ως προς τα όσα βλέπω στο έγγραφο, αλλά ως πρώτη ανταπόκριση είναι αρκετά καλό. Αλλά θα ήθελα πιο συγκεκριμένα από τα αποτελέσματα, πιο καλή και συγκεκριμένη πρόοδο και βέβαια ενημέρωση εν μεταξύ. Ευχαριστώ κύριε Κέλλας. Ευχαριστώ και θα συμφωνήσω και εγώ ότι χρειαζόμαστε πιο πολλά στοιχεία συγκεκριμένα. Ευχαριστώ όλους όσοι ήρθαν για να μας ενημερώσουν. Ιδιαίτερα για την Κολομβία λοιπόν. Μας μιλήσατε για τα τρία τελευταία χρόνια. Εμείς καταθέσαμε ένα αίτημα το καλοκαίρι μόλις, το σε ένα οδικό χάρτη, ένα φύλλο πορείας που θα σας καθοδηγούσε για το μέλλον, για να βλέπουμε προς τα που τίνεται. Επομένως, το να στρέφουμε το βλέμμα συνέχεια προς το παρελθόν δεν βοηθάει τόσο πολύ. Πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα προς το μέλλον. Και πολύ καλά όλα αυτά τα οποία κάνατε στο παρελθόν, αλλά το να υποδεχθείτε αντιπροσωπείε τη Amnesty International, τη Διεθνού Αμνηστία ή να τηρείτε τι ε, διεθνεί συνθήκε, όσο καλό και να είναι, δεν σημαίνει και κανένα καταπληκτικό κατόρθωμα, γιατί είναι κάτι το αυτονόητο. Ερωτώ λοιπόν πώ μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, πώ μπορούμε να ενημερωθούμε για το τι σκοπεύετε να κάνετε από εδώ και μπρο. Ποιο είναι το φιλοπορία, σε πάση περιπτώσει, για εσά. Για δε το Περού, λέτε στο έγγραφό σα ότι αποτελεί μια επισκόπηση των ε, ε, προτάσεων θεσμικών, ε, πολιτικών κτλ. Φύλλο πορείας όμως δεν βλέπουμε. Πότε μπορούμε να το δούμε. Αυτή είναι η ερώτηση για το Περού. Συμφωνώ με τον ε, Μπεντ Λάγκ ότι πρέπει να αναλύσουμε πολύ προσεκτικά τα έγγραφα αυτά. Χρόνο δεν έχουμε αρκετό βέβαια μέχρι τις ψηφοφορίες τώρα το απόγευμα. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε. Πότε θα ακούσουμε τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που αναφερθήκατε στις οργανώσεις Ψηφοφορία δεν θα έχουμε στις το απόγευμα. Α, όχι. Σχόλια εκτός μικροφώνου δυστυχώς δεν μεταφράζονται. Καλά, ε, έστω, μέχρι τις 27 του μηνός πώς θα τα καταφέρουμε όλα αυτά. Θα προλάβουμε να δούμε όλους αυτούς τους εκπροσώπους. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, γιατί θέλουμε να δούμε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και όχι μόνο τις κυβερνήσεις. Αν καταφέρουμε μέχρι τις 27 του μηνός, θα είμαι πολύ ευτυχή. Αλλά επιμένω, όπω είπα, να δούμε αυτούς τους εκπροσώπους και να ενημερωθούμε συγκεκριμένα για το φιλοπορίας, για τα φύλλα πορείας. Ευχαριστώ. Μέχρι την ψηφορία προβλέπεται για τις 26 και 27 Νοεμβρίου έχουμε τη δυνατότητα. Εάν ο Μάριο Νταβίτ και ο Μπερτ Λάγκε το επιθυμούν ε, να γίνει μια συνεδρία είτε της ε, ομάδας για την υλοποίηση, της ομάδας εποπτείας. Θα είναι σύντομη βέβαια για να μελετηθούν, να αναλυθούν τα έγγραφα των δύο κρατών. Ενδεχομένως δε και να συναντηθούμε με άλλους εκπροσώπους. Αλλά αυτό θα είναι δίκη σας πρωτοβουλία. Κύριο Σόλτς, ευχαριστώ και εγώ υποστηρίζω την πρόταση αυτή. Δηλαδή μέχρι τις 27 του μήνος να αξιοποιήσουμε το χρόνο που θα έχουμε. Ευχαριστώ πολύ τους ε, τους προσβευτές που ήρθαν να μας επισκεφθούν. Και σημειώνω ότι έχουμε συζητήσει επί δύο μισή χρόνια το αν είναι μισοάδιο ή μισογεμάτο το ποτήρι. Και δεν έχω ακόμη πιστεί ότι είναι μισογεμάτο. Από την ανάγνωση των αγράφων. γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει αυτό το φύλλο να περιγράφει συγκεκριμένα μέτρα δεσμευτικά, δραστηριότητε που θα οδηγήσουν στην αλλαγή τη κατάσταση. και έτσι ναι μεν σημειώνω ότι έχετε επιτύχει κάποια πρόοδο και στο γραπτό κείμενο μας επισημαίνεται βελτίωση της κατάστασης αλλά, αλλά ταυτόχρονα έχουμε προβλήματα ίσως ε, αυτονόητα λίγο πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει και εμείς να εξηγήσουμε τι κάνουμε, τι κάνετε για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, να βελτιωθεί και ως εκ τούτου χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια. Βλέπω λοιπόν εδώ υποχρεώσεις στο έγγραφο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τις εργασιακές σχέσεις κτλ. Αν όμως συγκρίνουμε τα διαγραφά αφενός, δηλαδή αυτό που αφορά το, τις δικές μας σχέσεις αφετέρου, δε εκείνο που αφορά τις σχέσεις της Κολομβίας με τις ΗΠΑ, το οποίο είναι πολύ πιο σαφές, βλέπουμε ότι πολλά ακόμα μένουν να γίνουν στη σχέση, μας, στη σχέση σας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνουμε ότι σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο και άλλοι εταίροι σας ε, απαιτούν ή προάγουν ή ζητούν ένα πλαίσιο για τη βέλτιση της κατάστασης. Ίσως θα ήταν καλό να αναλύσουμε το έγραφό σαφέστερα. Συμφωνούμε να οργανώσουμε λοιπόν εις βάθος συζητήσεις μέχρι τις συνεδρίες της 26ης-27ης. Βεβαίως θα προσκληθούν εκπρόσωποι των δύο κρατών στη συνεδρίαση. Ο Μάριο για να κλείσουμε. Κύριε Πρόεδρε, μου φαίνεται παίρνοντα δεδομένο ότι θα έχουμε τέτοιου είδου συνάντηση. Αυτό εξαρτάται από το πρόγραμμά μα. Γιατί πρέπει να σα υπενθυμίσω ότι κάναμε ήδη μια ακρόαση στην Επιτροπή μα. Πολλέ ε, ακροάσει από διάφορε ομάδε οργανώθηκαν. Ε, υπήρχε επίσης ε, και στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων μια ακρόαση. Την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο ήρθαν τα συνδικάτα και μας επισκέφθηκαν. Βεβαίω ευχαρίστω, είμαστε πάντοτε ανοιχτοί στη συζήτηση, αλλά αρκεί να μην αλλάξουμε την προθεσμία τη 26ης, 27ης, γιατί έχουμε και τις εποπτικέ ομάδες, οι οποίες επίσης ε, μπορεί να ε, το συζητήσουν αυτό πριν από την συνεδρίαση στην οποία αναφέρεστε. Πάση περιπτώσει, το λέω αυτό ενημερωτικά. Και δεν νομίζω ότι όλες αυτές οι ώρες αυτές οι ακροα αλλάζουν και τίποτε επί τη ουσία να σα πω την αλήθεια. Merci infiniment. Merci. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Το απόγευμα ο Ρόμπερτ Μίτσομς Στέρντι θα προεδρεύσει της Επιτροπής μας. Γεια σας και καλή όρεξη.